Παρακαλώ καθίστε. Μπορούμε να αρχίσουμε σχεδόν στην ώρα μας, έστω και αν ε, τα έδρανα δεν είναι ακόμα γεμάτα. Αλλά σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο μας ε, και τον ε, Υπουργό, ο οποίος ήταν ακριβέστατος. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό και τη χώρα του για την ε, τεράστιες ε, πρόοδους που έχουν επιτευχθεί, αυτή η τεράστια μεταρρύθμιση που έγινε με ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε θέματα ασφαλείας, ε, κράτους δικαίου και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς όμως διαπιστώσαμε, ελπίζουμε όμως αυτό να το αναιρέσουμε σε μια επόμενη φάση, όσον αφορά στην ε, governance, ε, δηλαδή τη διαχείριση του κράτους, την καταπολέμηση της, ανεργίας, ε, της διαφθοράς όλα αυτά έχουν μεν προχωρήσει αλλά χρειάζονται ακόμη βελτίωση. Για το θέμα των ε, θεωρήσεων, της βίζας. Αυτό το θέμα ε, έβαζε την Αλβανία στην ίδια κατηγορία με την ε, Σερβία, την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρόοδοι είπαμε όμως έχουν γίνει η πολιτική επικαιρότητα της ε, χώρας ταράχθηκε ιδιαίτερα από τις αντιθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης για το θέμα των εκλογών. Ακόμη βέβαια δεν έχει λυθεί αυτή η διαφορά και δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε μια πραγματική πολιτική μεταρρυθμίσεων. Αυτό το σενάριο υποσκάπτει και τις ε, και τη συνέχεια που θα πρέπει να δώσουμε στο μέλλον. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, εσείς να μας τα πείτε καλύτερα, να σας ακούσουμε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κι εμείς μια καλύτερη άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Πρόεδρε κύριε Αλμπερτίνη αξιότιμα μέλη ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι χαρά μου να έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι νόπιό σας δύο εβδομάδες μόνο μετά α, την απάντηση του Πρωθυπουργού Μπερίσα στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Επίτροπο Φίλε. Με μεγάλη υπευθυνότητα και επαγγελματισμό ε, προετοιμάστηκε η απάντηση αυτή με, από τη διοίκησή μας ε, και πολύτιμη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ομάδων συμφερόντων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου επίσης δεσμευτήκαμε και εμείς να ε, κάνουμε αυτά που ε, έλεγε το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και για τη χώρα μας και για τους πολίτες από πλευρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κάποτε είμαστε η πιο απομονωμένη χώρα στην Ευρώπη και τώρα επίκειται ε, σημαντική απόφαση να ληφθεί για να έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν στο Σέγγεν χωρίς ε, βίζα οι πολίτες μας. Το όνειρό μας αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Στα πλαίσια αυτά Έχω την ευκαιρία και θα ήθελα να σα εκφράσω τη βαθιά μας ε, γνωμοσύνη προς εσά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στεναρή υποστήριξη και την ε, ενθάρρυνση να πληρώσουμε όλα τα απαραίτητα κριτήρια που τελικά θα οδηγήσουν στην απόφαση να αρθεί σύντομα επίση και για την Αλβανία το καθεστώς θεώρησης. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμα σημαντικότερο τώρα ο ρόλο σα και ε, εκ των όνου Κάνευ με τη θέση ισχύ τη Λισαβόνα, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αναγνωρίζω ότι η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για μας αλλά και για σας ως εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένε από τις πρόοδους και τα επιτεύγματά μας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα σας έχουν ενημερώσει και θα σας ενημερώσουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, τα benchmarks. Ε, μερικοί από εσά τα γνωρίζετε ήδη, διότι Έχετε μεταβεί στην Αλβανία πρόσφατα και είχατε την ευκαιρία να τα διαπιστώσετε ήδη. Έχει κάνει σημαντική ε, πρόοδο η Αλβανία για την ασφάλεια. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πάνω από 600.000 βιομετρικά ε, διαβατήρια και πάνω από 2 εκατομμύρια ταυτότητες αστυνομικές σε ένα πολύ σύντομο διάστημα. Κάθε πολίτης είναι γραμμένο σε δηματολόγιο και έχει ένα μόνιμο αριθμό, προσωπικό αριθμό μητρό. Έχει κάνει σημαντικές πρόοδους επίσης ε, στα σύνορα, στη φύλαξη των σύνορων, στο άσυλο και στη μετανάστευση η χώρα. Έχουμε βάλει στα σύνορά μας τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και βιομετρικούς ε, ε, μετρητές. εκπαιδεύουμε αστυνομικούς έχουμε στρατηγική και πρόγραμμα εθνικό, πράγμα που οδήγησε σε ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων μας. Πλήρως συνεργαζόμαστε για να πληρώσουμε ε, τις θήκες και τα κριτήρια ένταξης. Στο τρίτο μπλοκ ε, για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια έχουμε αυξήσει τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της εγκληματικότητας, του τράφικινγκ. Ε, έχουν εγκριθεί πολύ σημαντικοί νόμοι και θα ήθελα εδώ να αναφέρω το ε, νόμο για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, το λεγόμενο νόμο ε, κατά της μαφίας, για να ε, περιορίσει ε, την εγκληματική δραστηριότητα ομάδων ή ατόμων. Επίσης έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την πρόληψη της διαφθοράς και για τη διακυβέρνηση με διαφάνεια και τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις ε, διαφθοράς που διώκονται και μεταξύ αυτών και ψηλοί αξιωματούχοι. Έχει μάλιστα αρθεί και ασυλία δικαστών. Η εφαρμογή λοιπόν της αντίστοιχης ε, νομοθεσίας και το πρόγραμμα δράσης κατά ε, του τράφικινγκ των ναρκωτικών και τα λοιπά συνεχίζεται. Και έχει μειωθεί πολύ το φαινόμενο αυτό. Είναι πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου για αυτά τα θέματα. Ε, τα βασικά στοιχεία όμως για την επιτυχή εφαρμογή είναι η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα. Στο τέταρτο μπλοκ, το Εθνικό ε, Σχέδιο Δράσης για την συμπερίληψη των Ρωμά επίσης έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται. Προστασία ε, από διακρίσεις έχει γίνει νόμος και είναι πολύ σημαντικό ως εξέλιξη και αυτό και ο Επίτροπος ε, είναι μια θέση που εγκρίθηκε από την Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, Επίτροπο για την Άση των Διακρίσεων και για την Ισότητα και προσεχώ θα διοριστεί από το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την ευθύρια τη ε, έκφραση, η Βουλή τη ε, Αλβανική Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε έγκριση νόμων κατά της συγκοφαντικής δυσφήμισης. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τώρα, είμαστε πιο κοντά σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς. Οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα, προβλεψιμότητα ε, είναι εγγυημένα και έχουν διατηρηθεί ε, εξάρτητα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πέρυσι είχαμε θετική επίσης ε, οικονομική εξέλιξη και έδειξε αυτό ότι η οικονομία μας είναι αισιόδοξη και δυναμική. 3,3% ήταν η μεγέθυνση της οικοδομίας το 2009. Επενδύουμε ε, στην ενέργεια και στις διασυνδέσεις γενναία και ενεργά, καθώς θέλουμε να είμαστε σημαντικός περιφερειακός παράγων στην ενέργεια. Το ίδιο μπορεί να υποθεί και για την υποδομή των ε, αυτοκινητοδρόμων έχει ε, αυξηθεί με στρατηγικό στόχο να συνδέεται με περιφερειακές αγορές και χώρες καλά και ευρύτερα η Αλβανία. Αυτό είναι το όραμά μας για την περιφερειακή εξωτερική πολιτική όπου η ε, Αλβανία ε, διαδραματίζει ένα ρόλο σταθεροποιητικό ευημερίας και ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνο μεταξύ επικοινωνίας παντού και αυξημένων ε, ανταλλαγών και συναλλαγών μεταξύ των λαών, το πολιτισμό, της οικονομίας, του πανεπιστημίου, της κοινωνίας των πολιτών, των μίντια, θα γνωρίσουμε ένας καλύτερα τον άλλον και θα υπερβούμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Εξαιρετικές είναι οι σχέσεις με όλους τους γείτονές της και με όλες τις χώρες της περιοχής. Και ε, βεβαίως βελτιώνονται οι σχέσεις με τη Σερβία, διότι θεωρούμε ότι η περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση είναι εκ των ουκάνευ για να ε, επιταχυνθεί η ολοκλήρωση και ένταξη όλης της περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας. Γνωρίζουμε τις ε, ισχυρές μας πλευρές, αλλά ξέρουμε και τα προβλήματά μας. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι, θα πρέπει να συνεργαστούμε σκληρά ε, για να ανταποκριθούμε στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει, και, συγγνώμη, η κυβέρνηση την πεποίθησή της και τη δέσμευσή της ε, ότι θα παρακολουθήσει και θα συνεργάζεται και με την αντιπολίτευση ε, για την προσπάθεια αυτή, για να υπερβούμε τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Η πλειοψηφία κάλυσε λοιπόν τη αντιπολίτευση ε, σε ένα επικοδομητικό διάλογο ε, δύο βασικούς γνώμονες, τη διαφάνεια και το σεβασμό ε, του συντάγματος της χώρας. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση πρότεινε στην αντιπολίτευση την Προεδρία και την πλειοψηφία σε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Επίσης προτείναμε να συσταθεί ένα σώμα διοκτών εισαγγελέων για να ε, εξεταστούν όλες οι αιτιάσεις αντιπολίτευσης. Η χώρα είναι δημοκρατική και ευρωπαϊκή, μέλος του ΝΑΤΟ και προτίθεται να γίνει και μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σεβόμαστε το Σύνταγμα και ε, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που θα πρέπει να είναι δεδομένη. Ε, το Αλβανικό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να ανατρέψουν δικαστικές αποφάσεις κυβέρνηση είναι πρόθυμη να ε, ακούσει ε, τις αιτιάσεις της ε, αντιπολίτευσης, να απευθυνθούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο και στην Λόγο Επιτροπή και θα δούμε τι θα προκύψει. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου που κάνει τώρα το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν εγγράφεται στο πλαίσιο του σεβασμού της δημοκρατίας και έχει και αρνητική επίδραση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και στην ευρωπαϊκή μας πορεία και ατζέντα. Επίσης, προσφέραμε στην αντιπολίτευση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου για τις ερχόμενες εκλογές ε, βάσει των όσων μας ζητάει ο ΑΣΕ και ο ΔΙΡ. Θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να καλεί και να εργάζεται προς ένα επικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος να προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή μας ολοκλήρωση, ένταξη και είναι εθνικός αυτός ο στόχος για όλους τους Αλβανούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο, εισηγητής της Αλβανίας, για την Αλβανία. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κύριο Μέτα. Δεν θέλω να υποβάλω ερωτήματα καθώς πρόσφατα ε, επισκέφτηκα στα πλαίσια του ρόλου της σύνταξης της έκθεσης για την Αλβανία τη χώρα και επομένως εκεί συζήτησα αναλυτικά με τους εκπροσώπους, ε, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών έχω μια καθαρή εικόνα. Θα συζητήσουμε το, ε, την έκθεση στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Θέλω να συμφωνήσω με τα, αυτά που είπε ο κύριος Μέτα, ότι πράγματι έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία και αυτά πρέπει να τα χαιρετήσουμε. Ε, νομίζω ότι η προπτική στην οποία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη της ένταξης της Αλβανίας και των δυτικών Βαλκανίων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πράγματι ένα κίνητρο για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, για να βελτιωθεί το επίπεδο, για να λυθούν μια σειρά προβλήματα. Αυτό το κίνητρο παραμένει ζωντανό μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και της αλβανικής κοινωνίας και επομένως από τη δική μας την πλευρά, την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών, <clears throat> ειδικά για μας από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πέρα από τις υποδείξεις, τις παρατηρήσεις τι άλλο πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί αυτό το θέμα. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι και το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο ως ελεκτή το τι δεν κάνει και τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά ως αρρωγού σε μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει και που θα είναι προς το καλό της περιοχής και προς το καλό του λαού της Αλβανίας. Η παρατήρησή μου είναι ότι η πολιτική σημερινή κατάσταση που είναι δύσκολη και αδιέξοδη <clears throat> είναι πολύ κρίσιμο θέμα στην πρόθεση και των ε, άλλων μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Εκεί υπάρχει μια αδιέξοδη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο καθώς το Κοινοβούλιο στην ουσία δεν λειτουργεί, ε, ο διάλογος είναι αλυσιτελής, δεν βγάζει αποτέλεσμα, δεν φαίνεται διέξοδος. Προφανώς υπάρχουν πολιτικές ε, αιμονές οι οποίες ε, δεν ε, βλέπω πώς αλλιώς μπορούν να λύνουν παρά σε σεβασμό στη λαϊκή εντολή, στο συνταγματικό πλαίσιο και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Ε, ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί λύση, ούτως ώστε η κατάσταση όσο αφορά αυτό το επίπεδο να ομαλοποιηθεί και να μπορέσει να συγκεντρωθεί η προσοχή των πολιτικών δυνάμεων της αλβανικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η τελευταία μου παρατήρηση, συμφωνώ με αυτά που ανέφερε ο κύριος Μέτα, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο κράτος δικαίου, έχουν ψηφιστεί σημαντικότατοι νόμοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της διαφθοράς, της ε, ε, τράφικινγκ, εμπορίας ναρκωτικών δικαιωμάτων. Το κρίσιμο θέμα που πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της, νομίζω, η αλβανική κυβέρνηση και οι αλβανικές ε, δυνάμεις είναι στην εφαρμογή. Και η εφαρμογή είναι μια δύσκολη υπόθεση και εκεί ακριβώς ε, τελειώνω με αυτή την παρατήρηση ε, ε, να συγκεντρώσουμε και εμείς την προσοχή μας αν όπως είπα στην αρχή η δική μας η προσπάθεια θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε όχι μόνο να τσεκάρουμε και να ελέγχουμε προκειμένου αυτά τα πράγματα και στην πράξη να αντιμετωπιστούν. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Ο, κύριος Κούκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Συγχαρητήρια και σε εσά και για τη χώρα σας για δύο ουσιαστικά πράγματα. Πρώτον, το ότι απαντήσατε στο ερωτηματολόγιο το προενταξιακό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεύτερον, συγχαρητήρια για την πρόοδο που έχετε σημειώσει όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Πήγα πρόσφατα στην Αλβανία και είδα επί τόπου ότι τα πράγματα λειτουργούν και ότι η τεχνική διάσταση, αν θέλετε, όλων αυτών των ζητημάτων λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς πολιτικής στο δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το εφιστάμενο πολιτικό διέξοδο στο Αλβανικό Κοινοβουλίο, όπου ουσιαστικά η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει τον δρόμο της Αλβανίας, την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια νομοθετήματα τα οποία πρέπει να εγκρίνει η Αλβανία προκειμένου να πετύχει την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάμεσα στα νομοθετήματα αυτά χρειάζεστε, και για τα νομοθετήματα αυτά χρειάζεστε και την υποστήριξη αντιπολίτευσης. Πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό. Βεβαίως πιστεύω ότι ε, όσο συντομότερα λυθούν τα πολιτικά προβλήματα τόσο το καλύτερο για τη χώρα και θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών και ότι οι αποφέσεις των θεσμών αυτών θα πρέπει να τύχουν σεβασμού, να τηρηθούν από όλους, όλους τους πολιτικούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η πρώτη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Νομίζω ότι θα αποτελεί αυτό μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα μέλη του Αλβανικού Κοινοβουλίου καθότι θα κληθούν να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί εδώ πέρα στις Βρυξέλλες από ό,τι ουσιαστικά στην χώρα τους. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταφέρουν να επιβιώσουν εδώ στις Βρυξέλλες, να καταφέρουν να περάσουν μαζί όλες αυτές τις ώρες ε, και για τη συζήτηση και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος και του ε, δείπνου. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο ζήτημα της ε, περιφερειακής ανάπτυξης, να συγχαρώ την χώρα σας για τον τομέα αυτό. Ξέρω ότι έχετε καταργήσει το καθεστώς θεωρήσεων για τις περισσότερες χώρες της ε, περιοχής σας, τις όμορες χώρες της ε, Αλβανίας και θα ήθελα να δω και ανάλογες τέτοιες ε, δραστηριότητες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούκκινο, κύριος Δανζόν, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, την Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας και την εργασία της κυβέρνησής σας σε όλους τους τομείς. Είναι διαμφισβήτητες οι πρόοδοι που έχετε πράξει. Η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο και καθιστά αυτό το μποϊκότ της αντιπολίτευσης προς το Κοινοβούλιο πραγματικά ανεύθυνη. Ο κύριος Κούκεν ανέφερε κάτι στο τελευταίο σημείο που αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Η κυβέρνησή σας και εσείς παίζεται ένα ρόλο πολύ σημαντικό σε αυτή την περιοχή που είναι μια δύσκολη περιοχή παρόλα αυτά για να, να προσφέρετε προπτικές για το μέλλον. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι έγινε στην επίσκεψή σας που πήγατε στη Σερβία. Θα ήθελα επίσης να ξέρω τι γίνεται και με την ε, πρώην ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας όπου λέγεται ότι οι Αλβανοί της ε, Φιρόμ βιώνουν άσχημα την κατάσταση και θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε εσείς για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ναζό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μέτα, έχετε το λόγο, 5-6 λεπτά για απάντηση. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω αυτή τη στιγμή και να μιλήσω πάρα πολύ για τις πρόσφατες εκλογές, απλώς θα πω μερικά πράγματα. Για πρώτη φορά σε περίοδο 20 ετών, ο εκλογικός κώδικας καθώς επίσης και η νομοθεσία και η ύπατη επιτροπή για τις εκλογές ουσιαστικά σχεδιάστηκαν από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον κύριο Ράμα. Και ουσιαστικά εμείς εγκρίναμε όλα αυτά τα οποία πρότεινε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω πράγματα που έχουν υποθεί. Οι εκλογές αυτές ήταν πάρα πολύ καλές από νομικής πλευράς και από τεχνολογικής όμως πλευράς. Το είπε και ο ΑΣΕ. Καταφέραμε να καταγράψουμε κάθε ψήφο σε κάθε εκλογικό γραφείο της χώρας. Τα δύο βασικά κόμματα είχαν ίση αντιπροσώπευση στην διοικητική διαδικασία, 50% και 50% για τα δύο βασικά κόμματα. Και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουν επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα αυτά για το σύνολο της χώρας. Τώρα λένε ότι θέλουν να κάνουν κάποιε έρευνε όσον αφορά τι πρόσφατε αυτέ εκλογέ και έχουν αφαιρθεί σε διάφορα ζητήματα. Και η πλειοψηφία κάνει ό,τι μπορεί. Του έχουμε προσφέρει κάθε δυνατότητα. και εμείς ως πλειοψηφία τους κάναμε πάρα πολλές παραχωρήσεις, να είναι επικεφαλή σε διάφορες επιτροπές, να ξεκινήσει μια εξεταστική επιτροπή. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αρχίσει να εργάζεται και από σήμερα ακόμα, αν το επιθυμούν. Για οποιαδήποτε αιτίασή τους, για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε αίτημά τους, εμείς ήμασταν ε, έτοιμοι να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Λένε τώρα ότι θέλουν να γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων. Υπήρχε όμως η επίσημη φορευτική επιτροπή και κάθε μέλος της έγινε αποδεκτό από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Λέμε λοιπόν ότι το αίτημά τους αυτό δεν είναι συνταγματικό γιατί ουσιαστικά βάλει κατά της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και βάλει κατά της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων της χώρας και έχει πάρει το Σταγματικό Δικαστήριο μια απόφαση στο παρελθόν που έχει να κάνει με τις ε, εξεταστικές αυτές κοινοβουλευτικές επιτροπές που μπορούν να εξετάσουν ε, σύμφωνα με την απόφαση αυτή τα πάντα, αλλά όχι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το κόμμα της αντιπολίτευσης όμως έχει διαφορετική γνώμη. Εμείς, ακόμα και σε αυτό, είμαστε ιδιαίτερα υποχρεωτική γιατί δεχτήκαμε μία πρόταση που κάνανε να απευθυνθούν στην Επιτροπή της Βενετίας, που δεν αποτελεί θεσμό βέβαια της χώρας μας, της Αλβανίας. Αποδεχθήκαμε όμως την πρότασή τους αυτή να πάνε στην Επιτροπή της Βενετίας, γιατί η Επιτροπή της Βενετίας μας είχε βοηθήσει στο παρελθόν με την σύνταξη του στάγματός μας. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει μια εξεταστική επιτροπή της εργασίας της σήμερα ή αύριο και να ερευνήσει διάφορα ζητήματα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα μας έχει πει ότι θα πάει είτε στο Θεγματικό Δικαστήριο είτε στην Επιτροπή της Βενετίας. Εμείς θα δούμε ποια είναι η γνωμοδότηση των σωμάτων αυτών και θα συμμορφωθούμε με τη γνωμοδότησή τους. Έτσι έχει η κατάσταση. Συμφωνώ με τις ε, ανησυχίες ορισμένων ευρωβουλευτών που ε, αναφέρθηκαν στο ότι θα πρέπει το Αλβανικό Κοινοβούλιο να περάσει με ενισχυμένη πλειοψηφία κάποιους νόμους. Ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αποτελεί μόνο η υποχρέωση και δέσμευση της ε, κυβέρνησής μας, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικά δέσμευση και της ε, αντιπολίτευσης. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εθνικό στόχος, όχι μόνο για την Αλβανία ως χώρα, αλλά και για τους Αλβανούς ως έθνος. Γιατί μόνο μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας και όλων των χρόνο που ζουν οι Αλβανοί θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους Αλβανούς να συσπηρωθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβιώσουν με όλους τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η αντιπολίτευση να αναλάβει τις ε, ευθύνες της και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ότι σήμερα που ο Πρωθυπουργό υπέβαλε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης προσωπικά είπε ότι θα πρέπει ο κόσμος να εξεγερθεί. Για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο, ποιο μήνυμα θέλει να στείλει. Ο ίδιος ο λαός της Αλβανίας έχει κουραστεί πια, έχει αγανακτήσει, έχει βαρεθεί να ακούει για μποϊκοτάρισμα, δεν θέλει να ακούει πλέον για απειλέ χρησιμοποίησης βίας και θεωρώ ότι το μήνυμα το οποίο στέλνει ο ηγέτης της αντιπολίτευση είναι λανθασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει στάση η αντιπολίτευση το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί τους προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούν όμως να θέτουν τη χώρα, τη σταθερότητα της χώρας και το κράτος δικαίου σε κατάσταση ομοιρίας και ουσιαστικά να υπονομεύουν το ίδιο το μέλλον της χώρας στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά δεσμεύομαι να κάνω κάθε τι το δυνατό και νομίζω ότι και η πλειοψηφία άλλωστε είναι απόλυτα δεσμευμένη. Θα πρέπει όμως από την άλλη να έχουμε και μια πιο υπεύθυνη και επικοδομητική στάση από την ε, αντιπολίτευση και μην ξεχνάνε ότι το εθνικό συμφέρον είναι πιο σημαντικό από το προσωπικό συμφέρον. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Αν όμως βάλουμε κατά της απόφαση του δικαστηρίου θα στείλουμε ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα για το σύνολο της χώρας θα λέμε ουσιαστικά ότι δεν σεβόμαστε το κράτος δικαίου, αλλά ότι οι αποφάσεις μας τελικά επηρεάζονται από τα προσωπικά πολιτικά συμφέροντα των πολιτικών της Αλβανίας. Όσον αφορά τώρα την ευρύτερη περιοχή, σαφώς θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες, με όλους τους γειτονές μας. Και για αυτό το λόγο πήγα πρόσφατα στην Σερβία σε μια επίσημη επίσκεψη. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους Σαφώς οι απόψεις μας διείστανται όσον αφορά το καθεστώς του κοσυφοπεδίου. Συμφωνούμε πάντως ότι και το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να αποτελέσει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η διμερή συνεργασία για την σταθερότητα της γενικότερης περιοχής μας και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τόσο της Αλβανίας όσο και της Σερβίας όσο και της γενικότερης περιοχής. Και για αυτό το λόγο έχουμε δεσμευτεί να συνεργαστούμε περισσότερο και με τη Σερβία και να σημειωθεί πρόοδος γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και για αυτό το λόγο άλλωστε μονομερός καταργήσαμε την απέτηση θεώρησης για τους πολίτες της Σερβίας και ελπίζουμε ότι η ανάλογη απόφαση θα ληφθεί και από την κυβέρνηση της Σερβίας σύντομα. Προσπαθούμε επίσης να αυξήσουμε την περιφερειακή συνεργασία ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό για όλη την περιοχή. Πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας και να στονιστούμε καλύτερα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα βοηθήσει βασικά και την εικόνα και την αξιοπιστία της περιοχής μας. Τη στιγμή που ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στήσουν το ζήτημα της ε, ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων, καθώς επίσης και άλλες πτυχές της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περιοχής μας. Τώρα όσον αφορά την ε, Μακεδονία, λέει ο μιλητής, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα καλύτερο κλίμα. Θα θέλαμε να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος και να εφαρμοστεί η συμφωνία του ΟΡΙΤ Θέλουμε να εφαρμοστεί η Συμφωνία της Αχρίδας και θέλουμε να βελτιωθούν οι σχέσεις της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ζητάμε από την αλβανική κοινότητα και τους αλβανούς ηγέτες να δείξουν επικοδομητική στάση, να είναι υπομονετικοί και να εργαστούν στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων της χώρας αυτής. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Δίγεν, για τρία λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Μέτα, στην Επιτροπή μας. Ε, η ανταλλαγή αυτή απόψε είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την πρόοδο που έχει κάνει η κυβέρνησή σας και η Ελβανία πρόσφατα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε επιτυχές βήμα για οποιαδήποτε χώρα της περιοχής βελτιώνει τις εξελίξεις και στις άλλες χώρες. Βεβαίως κάθε χώρα αξιολογείται ξεχωριστά, μονομένα, αλλά συχνά βλέπουμε ολόκληρη την περιοχή ως ένα σύνολο. Και όταν κάτι πάει καλά σε μια χώρα, αυτό βοηθάει και τις υπόλοιπες και βελτιώνει και τις σχέσεις με τους γείτονες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Και βοηθούν και τη δική σας χώρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Φέτος, έστω και αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, η Αλβανία θα ενταχθεί στο σύστημα απελευθέρωσης από τις θεωρήσεις και γνωρίζοντας τι έχει προηγηθεί για άλλες χώρες ε, ως διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα φέρει μεγάλη αισιοδοξία ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα σας. Και θα παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε αυτή την αισιοδοξία του λαού για να ενισχύσετε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να επιταχύνετε και την ευρωπαϊκή σας πορεία προς την ένταξη. Ωστόσο, πάλι, θα πρέπει να πούμε και να λάβουμε υπόψη ότι οι προετοιμασίε για την ένταξη δεν είναι μόνο διοικητική φύσεως, είναι και πολιτικής. Και οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει, όλοι οι πολίτες της χώρας, θα πρέπει να υποστηρίξει ο λαός της χώρας, λέω και η κυβέρνηση, στις εξελίξεις. Μετά τις εκλογές είδαμε ανισχυτικέ ε, καταστάσεις στην Αλβανία. Αναφερθήκατε εκτενώς σε αυτά. Αν ήταν όμως σήμερα εδώ κύριος Ράμα στη θέση σας, άλλο θα μας έλεγε. Και πολύ πιστικά εξίσου για την κατάσταση. Οπότε εμείς δεν είμαστε εδώ βεβαίως για να αναμειχθούμε στα εσωτερικά σας, αλλά θα θέλαμε να λυθεί το πρόβλημα, τα προβλήματα. Και όταν υπάρχουν τέτοιες ε, αντιφατικές ε, δηλώσεις, δεν φταίει πάντα ένας και μόνο έτσι. Ελπίζουμε και οι δύο πλευρές να κάνουν κάποιους συμβιβασμού και βήματα έτσι ώστε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο να σπάσει το συντομότερο. Υπό την έννοια αυτή, θα ήθελα να σας ζητήσω ε, παρακαλώ να επεκταθείτε λίγο περισσότερο σε αυτό. Πώς βλέπετε τώρα τα επόμενα βήματα. Γιατί αν δούμε την ε, συμπολίτευση και την αντιπολίτευση ε, να εμένουν στις τάσεις τους και να μην κινούνται καθόλου. Ε, εσείς πώς αξιολογείτε τις μελλοντικέ εξελίξεις, γιατί είναι και πάλι πολύ ανησυχητικό και αν συνεχίσει θα είναι εις βάρος των πιθανότητων ένταξής σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Πακ, που είναι σκεώδης εισηγήτρια για την Αλβανία εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών ε, που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Την τελευταία δεκαετία έχουμε ειδωθεί πολύ συχνά. Σας έχουμε δει πρωθυπουργό, σας έχουμε δει εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης και τώρα στην τελευταία συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία σας είδαμε να ε, καταπολεμείτε με μεγάλο ζήλο ε, τον εκλογικό νόμο τότε Ράμα Μπερίσα. Τώρα το δεχτήκατε. Δεχτήκατε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί τότε για τον εκλογικό νόμο και ένας που εργάστηκε για τον νόμο αυτό Τώρα τα έχει βάλει με τον νόμο λες και είναι ανεμόμυλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ότι υπάρχουν πράγματα που είναι τόσο σοβαρά και τόσο βαριά που μια ολόκληρη αντιπολίτευση μήνες ολόκληρους δεν πάει στο κοινοβούλιο. Και τώρα πάει σποραδικά που και που και όποτε θέλει ξαναφεύγει για να μην χάσει και την εντολή της. Και καλή είπατε και για κοινωνικές ταραχές. Και ε, πώς μπορεί ένα κόμμα να καλέσει τον κόσμο να βγει στους δρόμους όταν η κατάσταση έχει ως εξή. Έχει και κυβέρνηση χώρα που δεν είναι μονομερής, δεν είναι μονοκομματική, προέρχεται από διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς, είναι συνασπισμός και είναι κόμματα τα οποία ε, πάλευαν, αντιπάλευαν το ένα το άλλο αλλά τα βρήκαν τώρα για να βοηθήσουν την Αλβανία να πάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όπως είπατε αυτό είναι στόχος και καθήκον όλων, ακόμα και εκείνων που μετά τις εκλογές βρέθηκαν στην αντιπολίτευση. Από το 1991 παρακολουθώ άμεσα την κατάσταση στη ε, Αλβανία και μπορώ να επιβεβαιώσω και αυτά που είπατε και εσείς και ο ΑΣΕ και ο ΟΝΤΙΡ οι τελευταίες εκλογές ήταν οι καλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Αλβανία. Συμφώνησαν όλοι οι επίτροποι και οι παρατηρητές και λοιποί. Αλλά και ακόμα και αν υπάρχουν κατηγορίες και αιτιάσεις εκ των υστέρων θα πρέπει αυτές να γίνουν αρμοδίως. Ε, τα παράπονα, α πούμε. Εγώ μέχρι σήμερα δεν καταλαβαίνω. Ε, έστω ότι η αντιπολίτευση έχει δικαιολογημένες κατηγορίε. Γιατί δεν τα πάει αυτά στο Συνταγματικό Δικαστήριο ή στην Κεντρική Αφορευτική Επιτροπή. Δεν αποφασίζει το Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Αν έχουν ανοιχτεί οι κάλπε ή ξέρω εγώ αν υπάρξει πρόβλημα. Ε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κύριο Ράμα τι λέει. Ε, Μήπω είναι ανυπόστατα τα στοιχεία και κάνει τη φασαρία όλη αυτή για πολύ προσωπικά συμφέροντα ε, τότε να το πούμε και αυτό με το όνομά του. Εγώ δεν θέλω να ε, κατηγορήσω ή να ενοχοποιήσω κανέναν. Ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Εγώ περιγράφω στοιχεία και γεγονότα και θα παρακαλούσα όλους τους ε, να τα δουν και ως στοιχεία. Δεν είναι μονομερή, είναι γεγονότα καθημερινά τα διαπιστώνει κανείς στην Αλβανία και γνωρίζω από πολλές συζητήσει που έχω με το λαό της Αλβανίας ε, ότι δεν θέλει ο λαός ε, συνέχεια να διονύζεται αυτή η συζήτηση. Θέλει μια κυβέρνηση που να λειτουργεί. Και δύο ερωτήσεις. Στην έκθεση του κυρίου Χουντή λέει ότι δεν περιορίζεται το τράφικινγκ. Τι γίνεται με το εμπόριο γυναικών, οργάνων, κατα... Ε, πίεση, ε, παραβίαση των παιδικών δικαιωμάτων, κακοποίηση των παιδιών, γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Και τι γίνεται με τον νόμο ισότητα και πώς αυτό εφαρμόζεται. Βεβαίως και υπάρχουν οι νόμοι. Πώς εφαρμόζονται όμω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Βάγκελ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό της Αλβανίας ε, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Μέτα για τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και ελπίζω ε, οι επιτυχίες αυτές να ε, συνεχιστούν και να έχουν αίσιο πέρα στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοβουλευτική κρίση αυτόν τον καιρό στην Αλβανία είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι η μοναδική κρίση. Τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά, ε, το ίδιο σχέδιο σε όλες τις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Μόλις βγει μια κυβέρνηση ε, ακολουθεί διαφορετική στάση από εκείνη που είχε όταν ήταν αντιπολίτευση. Και τούμπαλιν. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό ούτε για το κοινοβούλιο, ούτε για τη φήμη και τη λειτουργία του κοινοβουλίου, ούτε για τη δημοκρατία την ίδια. Στο κοινοβούλιο αυτό, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν παίρνουμε θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Δεν είναι ο δικός μας ρόλος αυτό να αποφασίσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Μιλήσατε για την περιφερειακή σημασία που έχει η χώρα σας. Μπορεί να συνεισφέρει και πάρα πολύ η Αλβανία με την πολιτική της. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά που εκκρεμούν στη γειτονία σας και εδώ πρέπει και εμείς να γνωρίσουμε ότι μια σταθερή Αλβανία μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων. Θα ήθελα τέλος να πω ότι εγώ είμαι εκπρόσωπο των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρώ πολύ σημαντικό να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όλων των μειονοτήτων. Και εκείνων που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Και βεβαίως και τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Η κυρία Φέζα. Δημόσιες ελευθερίες, εισηγήτρια για τις θεωρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό κύριο Μέτα για ε, όλα αυτά που μας είπε για την εκτενή ενημέρωση για την πρόοδο της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση. Είχαμε επανειλημμένα την ευκαιρία να το συζητήσουμε μαζί σας αυτό το θέμα και όχι μόνο αυτό, ότι όλα τα θέματα, την απελευθέρωση, το θεωρήσω. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό για τις ε, εξαιρετικές πραγματικά πρόοδους που έχει κάνει η Αλβανία ε, στον τομέα αυτό. Είδαμε και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πάρα πολύ θετική. παρόλο που απομένουν ορισμένα θέματα σε εκκρεμότητα και έχετε ακόμα δουλειά μπροστά σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Σχετικά με την επιστροφή ε, Αλβανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα αυτό ε, των Αλβανών που επαναπατρίζονται και πρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία. Ε, πώς καταπολεμείτε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Μας είπατε ορισμένα στοιχεία ήδη ποιοι είναι οι στόχοι σας και πού θέλετε να φτάσετε, αλλά θα με διέφερε να ακούσω ε, τι συγκεκριμένα αποτελέσματα θέλετε να έχετε πετύχει πριν τον Ιούλιο. Μέχρι την επόμενη αποστολή στην Αλβανία. Για να έχουμε ενημέρωση ε, για την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα των θεωρήσεων και πώς είστε έτοιμοι να απελευθερωθούν θεωρήσεις. Εγώ επιθυμώ να μπει σε αυτό το σύστημα βέβαια το συντομότερο η Αλβανία, αλλά θεωρώ επίσης ότι μπάλα είναι στο δικό σας γήπεδο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιταχυθεί η διαδικασία αυτή, αλλά και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια και σοβαρή δουλειά ε, στη δική σας πλευρά. Για να προχωρήσει το συντομότερο αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαγιόν. Ο κύριος Ράουτσεκ τώρα, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρούτσεκ μάλλον, και σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών για την Αλβανία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις και θα ήθελα να σας θέσω και κάποιες ερωτήσεις. Να σας συγχαρώ και εσάς και τη χώρα σας για την πρόοδο που έχετε σημειώσει για τα επιτεύγματά σας, όχι τους τελευταίους μήνες, αλλά τελευταία χρόνια θα έλεγα. όσον αφορά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις οικονομικές, εσωτερικής πολιτικής και όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Είπατε ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απασχολεί, θα πρέπει να απασχολεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό έλεγα και εγώ όλα αυτά τελευταία χρόνια σε όλους τους αξιωματούχους της Αλβανίας, είτε πρόκειται, από το, είτε για το κόμμα της πλειοψηφίας, είτε πρόκειται για τα, για τα υπόλοιπα κόμματα. Το ζήτημα της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων πρέπει να απασχολεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Στα πλαίσια μια κοινοβουλευτική δημοκρατία θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μπλοκάρει και να μπλοκοτάρει κανεί εργασίε του Κοινοβουλίου. Γιατί στα πλαίσια μια κοινοβουλευτική δημοκρατία το Κοινοβούλιο είναι η καρδιά του πολιτικού συστήματο. Γίνονται εκλογέ, πολλέ φορέ ε, η εκλογική εκστρατεία είναι δύσκολη και πικρή, αλλά μετά το τέλος των εκλογών θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις σύσσωμα να εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να περνούν νόμους, να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω και περνάω σε κάποιες ερωτήσεις. Ερωτήσεις όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας. Όντως, έχετε κάνει μια απτή πρόοδο τελευταία χρόνια, μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και το 2009, ενώ όλη η Ευρώπη με την εξαίρεση της Πολωνίας βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, εσείς ως Αλβανία τα πήγατε καλά. Παρ' όλα αυτά, η Αλβανία αποτελεί μία από τις πιο φτωχές χώρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Και χρειάζεστε μία σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Ακόμα και αν δούμε τα πράγματα μακροοικονομικά, η Αλβανία έχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα, ένα έλλειμμα στο τομέα του εμπορίου και νομίζω ότι υπάρχει και ένα σημαντικό έλλειμμα της τάξης του 7% όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Είπατε εσείς ότι δεν επρόκειτο να Προχωρήστε σε μια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όντως δεν χρειάζεστε αυτή τη στιγμή χρήματα, αλλά σε δύο ή τρία χρόνια, αν επηρεαστείτε από τη γενικότερη οικονομική κρίση, από την κατάσταση στην Ελλάδα, από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, θεωρείτε ότι είναι σωστή η απόφαση σε αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πρέπει επίσης να βελτιώσετε και την κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλά ρυθμισμένη αγορά ακινήτων, να υπάρχει μια διαφάνεια και σταθερότητα προκειμένου να μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Έχει τεράστιες δυνατότητες η χώρα σας όσον αφορά τον τουρισμό, τις μεταφορές, όσον αφορά πολλούς άλλους επιχειρησιακούς κλάδους. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητάνε μία διαφανή, σταθερή κατάσταση. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι τι προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ράουτσεκ. Ο Υπουργός για να απαντήσει σε ένα δεκάλεπτο ή δυνατόν. So, ε, ε, Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τον κύριο Βιγγένιν, τον πολύ καλό μου φίλο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει στοιχεία αδιάσυστα και πιστικά ως προς ε, το ορθόν και την αξιοπιστία των πρόσφατων εκλογών. Και να έρθω εδώ Όποτε θέλετε με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να έρθω και στη σοσιαλιστική ομάδα όποτε μας καλέσετε. Μέχρι τώρα ένα παράδειγμα έχουν καταθέσει. Μία περίπτωση η οποία αποδεικνύει την αξιοπιστία του εκλογικού συστήματος. Κατέθεσαν ένα έγγραφο σε ένα χωριό που ήταν ε, άκυρο, ε, όπου οι εκπρόσωποι των σοσιαλιστών έφυγαν το πρωί από το εκλογικό τμήμα αλλά αυτό το έγγραφο δεν μετρήθηκε ε, ούτε από το εκλογικό τμήμα ούτε από την Εφορευτική Επιτροπή. Παρόλο που το έχει ζητήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το γνωρίζει αυτό και το εκλογικό τμήμα. Αν το είχαν μετρήσει, το Δημοκρατικό Κόμμα θα έβγαζε μία έδρα ε, παραπάνω και ε, αυτό ε, θα του έδινε την απόλυτη πλειοψηφία. Ακριβώς λοιπόν επειδή απερίφθη αυτό το έγγραφο που δεν ήταν σωστό, ε, είναι η απόδειξη ότι το σύστημα δούλεψε σωστά. Δεύτερον. Αν θέλει κάποιος να κάνει μια επαγγελματική εξέταση μέχρι και δίωξη όλων των περιπτώσεων, έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να δώσει και ε, ε, οικονομική στήριξη στον εισαγγελέα έτσι ώστε η εισαγγελία, που είναι τελείω ανεξάρτητο όργανο από την κυβέρνηση, έτσι, να συστήσει και ομάδα εργασία, μια task force εισαγγελέων που να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Με όλες τις περιπτώσεις που το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει παράπονα, καταγγελίε για τις εκλογές, για να διεκπεριωθεί αυτή η υπόθεση το συντομότερο. Και πάλι θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι είμαστε πρόθυμοι σήμερα και αύριο, όποτε θέλετε, να αρχίσουμε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή και να συζητήσουμε για τη σύνθεσή της. Είπαμε να έχει πλειοψηφία ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Να έχει και τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, όπως το ήθελε. Και να αρχίσουν να εξετάζουν ό,τι θέλουν. Τα πάντα. Και να σεβαστούμε ό,τι απόφαση λάβει το Συνταγματικό Δικαστήριο ή η Επιτροπή της Βενετίας ε, για το αν θα ξανανοίξουν οι κάλπες ή όχι. Βεβαίω δια της αρμοδίας οδού εφόσον το ζητήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα από τα όργανα αυτά. Τι άλλο να κάνουμε πια, εγώ δεν ξέρω. Έχει το δικαίωμα η αντιπολίτευση να, ε, είναι, να προεδρεύει σε πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές και σας είπα πρώτα απ' όλα θα έχουν τη δυνατότητα να προεδρεύουν και στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένταξη. Έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό να διαδραματίσουν στο Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα της χώρας. και ας έρθουν στην Επιτροπή αυτή να αντιμετωπίσουν για την κυβέρνηση και να καταθέσουν οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, ανησυχία, μέλημα έχουν, εν περιπτώσει, για την πορεία της χώρας. Τώρα, για το trafficking, το εμπόριο ε, ανθρωπίνων όντων, γυναίκες κλπ. Δεν θέλουμε μόνο να χαράξουμε στρατηγικές, αλλά και ουσιαστικά η κυβέρνηση της χώρας μας έχει λάβει θέση για οικονομική υποστήριξη μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εδώ ε, και, και, χρόνια συγγνώμη, εργάζονται για την αποκατάσταση των θυμάτων, ε, για την κοινωνική τους ένταξη, για την προστασία γυναικών, παιδιών κτλ. Και είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι σε αυτή την υπόθεση. Για τις μειονότητες στην περιοχή μας κάθε λαός κάπου είναι πλειοψηφία και κάπου αλλού είναι ε, ε, μειονότητα. Κάπου αλλού είναι πλειονότητα και κάπου είναι μειονότητα. Όλες οι κυβερνήσεις λοιπόν και όλοι οι λαοί αυτό που θέλουν είναι να χρησιμοποιούν τις ίδιες προδιαγραφές και στάνταρ για, που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σέβονται τις μειονότητες. Και εκεί λοιπόν ε, είναι πολύ προσιλωμένη η αλβανική κυβέρνηση για να σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το ίδιο ζητούμε και από τους άλλους για τις αλβανικές μειονότητες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το εξής, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την αλβανική κυβέρνηση. Να ενταχθεί πλήρως η σερβική μειονότητα στο κοσυβοπαίδιο. Έχουμε λάβει ε, και δράσεις και τη χρηματοδότηση 400.000 ευρώ έχουμε δώσει για προγράμματα υποδομών και κοινωνικά στην Κρασάνιτσα που ε, δημιουργήθηκε από το σχέδιο Αχτισάρι και οι περισσότερες επιτροπές ε, εκεί ανήκουν σε μειονότητες. Είχε πάει και ο Δήμαρχος ε, στα Τύρανα και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι η μόνη λύση για σταθεροποίηση, ειρήνευση της περιοχής και βελτίωση των ε, ε, σχέσεων μεταξύ των λαών. Also uh, Ένα άλλο τώρα που ε, θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ την Τάνια που μας βοηθάει στο θέμα της βίζας. Εργαζόμαστε πράγματι σε συγκεκριμένα προγράμματα για την επανένταξη ε, των επαναπατριζόμενων το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών για ε, επαγγελματική εκπαίδευση, για κατάρτιση και απασχόληση. Λειτουργεί επίσης και το κέντρο για τους επαναπατριζομένους, για τους παλινοστούντες Αλβανούς και συνεργαζόμαστε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την ένταξή τους και για τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Μέχρι τον Ιούλιο πιστεύω θα είμαστε σε θέση να σας αναφέρουμε ειδικέ συγκεκριμένε προόδους. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και κατ' εμέ, η Αλβανία έχει καλύψει όλα τα benchmarks σχεδόν, αλλά γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται σε ορισμένου τομεί συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων αυτών μπλοκ. Ακόμα και μετά την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Διότι αυτές είναι προκλήσεις μακροπρόθεσμης όπως και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κλπ. Και αυτή η περίπτωση. About the economic situation. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση. Νομίζω ότι η οικονομική κατάσταση είναι υποέλεγχο, είναι σταθερή. Έχουμε θετική οικονομική ανάπτυξη στην Αλβανία, το είπατε και αυτό και εσείς πέρυσι, και αυτό οφείλεται σε κάποιους βέβαια συγκεκριμένου λόγους. Δεν σημαίνει ότι είμαστε μια χώρα χωρίς προβλήματα. Έχουμε αντλήσει όμως τα απαραίτητα διδάγματα από την πικρή οικονομική κρίση του 1997 με το σύστημα των πυραμίδων τότε και έχουμε πάντα κατά νου την μακροοικονομική σταθερότητα. Επίσης το τραπεζικό μας σύστημα παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα και θα παρουσιάζει στο μέλλον. Και είμαστε βέβαια πεπισμένοι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια αριθμητικά μας στοιχεία και το κάνουμε. Ένα από τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι ότι παγώσαμε κάποιες δαπάνες προκειμένου να κρατήσουμε υπό έλεγχο τα πάντα και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευράς μακροοικονομικής όσον αφορά τη σταθερότητα της χώρας, είτε για το παρόν, είτε για το μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον. Και ξέρουμε βέβαια ότι το μέλλον της οικονομίας μας εξαρτάται από τους ξένους επενδυτές οι οποίοι έρχονται και θα έρχονται στο μέλλον και αρχίζουν ήδη να επενδύουν σημαντικά στη χώρα μας, στις υποδομές, στην ενέργεια, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς. Ξέρετε ότι ε, η Αλβανία γίνεται όλο και πιο σημαντική από στρατηγικής πλευράς για τους ξένους επενδυτές, χάρη στην πολύ καλή σχέση που έχουμε με τις όμορές μας χώρες και χάρη στι ε, βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει στις υποδομές μας που μας συνδέουν με τις ομόρες μας χώρες. Σας ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τρία λεπτά ο κύριος Στάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, 28 Απριλίου έχουμε σήμερα. Και πέρασαν 20 χρόνια που ζήτησε η Αλβανία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ σας συγχαίρω για όλα όσα κάνατε τα τελευταία χρόνια. Η κομμουνιστική κληρονομιά στην Αλβανία βάρινε ιδιαίτερα και θα πρέπει να καλύψετε τεράστια κενά. Εγώ δεν μιλάω για την απολευθέρωση των θεωρήσεων και τέτοια πράγματα. Εμείς ελπίζουμε ότι γρήγορα θα καταργηθούν οι βίζες για την Αλβανία. Και η κυρία Φαγιόν το ανέφερε αυτό. Και πολλοί όλοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα όμως να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε την περιφερειακή συνεργασία που για τα Βαλκάνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή τη διαδικασία πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στη διάσκεψη του Μπορντό που πρόθεσαν του, νο, συγγνώμη, που πρόθεσαν οι Κροάτες και οι Σλοβαίνοι. Πώς εκτιμάτε την προετοιμασία αυτής της διάσκεψης. Η Ισπανία είναι μεταξύ των οργανωτών. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα για να εμβαθύνουμε ακόμη παραπάνω σε αυτές τις σχέσεις. Και μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την περιφερειακή συνεργασία. Ε, ακούμε ότι ε, ο Έντι Ράμα έχει προβλήματα με το Σαλί Βερίτσα. Μα αυτοί οι δύο επικοινωνούν άμεσα ο ένας με τον άλλον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν συναντηθεί τους τελευταίους έξι μήνες ποτέ και αν ναι πόσο συχνά. Ευχαριστώ. Σβένσον. Tack så mycket, herr ordförande. Och tack Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πριν από 40 χρόνια πήγα στην Αλβανία, πήγα στα Τύρανα, και οι φοιτητές φώναζαν συνθήματα φωνάζαν για το Στάλιν, ένα κλίμα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Διότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγει κανείς από μια τέτοια κατάσταση και να ξεχάσει όλη αυτή την κληρονομιά που έχει πίσω του. Πρέπει να δούμε τις θετικές πλευρές της κατάστασης που αλλάζει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πρέπει ταυτόχρονα να πω ότι στην Αλβανία και σε άλλες χώρες υπήρξαν προβλήματα στον εκδημοκρατισμό, έγιναν εκλογές, θα ξαναγίνουν εκλογές, υπάρχουν διαμαρτυρίες και θα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί Όλοι μας ελπίζουμε σε βελτιώσεις για να γίνει και η Αλβανία κάποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Πακ. Πρέπει να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα για να πεγκλωβήσετε όλη αυτή τη χάλια κατάσταση με το σωματεμπόριο και με τα διάφορα στη διακίνηση των ανθρώπων. Η κυρία Κοπά για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, τον κύριο Μέτα. Και θα ήθελα μαζί με τους συναδέλφους μου να χαιρετήσω την πρόοδο που έκανε η Αλβανία όλα τα τελευταία χρόνια και τις σκληρές προσπάθειες του αλβανικού λαού ε, στον δρόμο για την Ευρώπη. Το θέμα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Ε, πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση με κάθε τρόπο γιατί η μη λειτουργία του Κοινοβουλίου δημιουργεί ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που η Αλβανία τον βρίσκει μπροστά τη στο δρόμο για την Ευρώπη κάθε στιγμή. Θα ήθελα να μιλήσω ειδικά για το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας, που νομίζω είναι κεντρικό. Είναι γνωστές οι προσπάθειες που έχει κάνει η Αλβανία το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με τη Σερβία αλλά να αναφερθώ και ειδικά στη συνάντηση των Πρωθυπουργών πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ελλάδας και Αλβανίας στην περιοχή των Πρεσπών, όπου συζήτησαν πρόσφατα τα περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής. Εκείνο το οποίο όμως ειδικά από την ελληνική πλευρά μας προβληματίζει είναι η δηλωμένη προσπάθεια της αλβανικής κυβέρνησης για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή του Δυραχείου, που είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από την ελληνοαλβανική μεθόριο. Το θέμα ε, της διαχείρισης, το θέμα των όρων ασφαλείας, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων είναι για μας ένα μεγάλο ερωτηματικό και θα ήθελα ε, τη γνώμη του Υπουργού πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κοπά, ο κύριος ε, Πρέντα για δύο λεπτά. Δεν χρειάζομαι τρία λεπτά για να τα πω όλα. Δύο ερωτήσεις έχω για τον ε, κύριο Μέτα. Τι θα γίνει στο μέλλον. για τον νόμο σχετικά με τη συμφωνία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο νόμος και πώς θα λειτουργήσει τώρα για την διαδικασία ενσωμάτωσης ποιος είναι υπεύθυνος εκεί μιλάμε για ένα κόμμα μιλάμε για όλη την πολιτική τάξη μιας χώρας ποιον θεωρούν οι πολίτες υπεύθυνοι για αυτά τα, υπεύθυνο για αυτά τα χάλια ε, ευχαριστώ κύριε Πρέντο Υπουργός για την τελική απάντηση So. About, uh, our... Uh, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τις χώρες περιοχής, ιδιαίτερα με τη Σερβία, θα ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με τη Σερβία Πολύ σύντομα θα υπογράψουμε συμφωνία επανεισδοχής και πολλές άλλες διμερείς συμφωνίες τους έχουμε προτείνει. Και όπως υπογράμμισα και προηγουμένως, η Αλβανία μονομερός ήρε την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων για Σέρβους που έρχονται στην Αλβανία και ελπίζω να ισχύσει το ίδιο και από πλευράς σερβικής κυβέρνησης για τον Μπούρντο για το Σαράγεβο και τις σχετικές διασκέψεις. Πρέπει να σας πω ότι είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία. Προήλθαν από τη Σλοβενία και την Κροατία. Πολύ καλό παράδειγμα για το πώς δύο χώρες στην περιφέρεια συνεργάζονται. Όχι μόνο για να ε, ξεπεράσουν οποιαδήποτε διένεξη του παρελθόντος, αλλά για να βοηθήσουν όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι υπήρξε πρόβλημα στον Πόρντο και όλοι θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ε, η Ισπανική ε, κυβέρνηση ελπίζω να φροντίσει να είναι όλοι παρόντες στο Σαράγεβο και να γίνει μια καλή διάσκεψη των χωρών της περιοχής και να δώσουμε και ένα πρώτο θετικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καθώς επίσης και θετικά μηνύματα να λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή μας καταφέραμε μόλις πριν από ένα μήνα να διοργανώσουμε στα Τύρανα μια πολύ επιτυχή υπουργική ε, διάσκεψη υπουργών εσωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης ήταν πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι ήταν παρόντες ο Υπουργό Εσωτερικών τη Σερβία και ο Υπουργό Εσωτερικών του Κωσοβοπεδίου στην ίδια υπουργική διάσκεψη. Θα ήθελα δεν να υπογραμμίσω ότι για μα είναι πολύ σημαντικό, καθώ και για όλου βεβαίω, να ε, είναι όλοι παρόντε στο Σαράγεβο. Ε, ανεξάρτητα από την εγγραφή. Δηλαδή, ή από την επικεφαλίδα. Θα πρέπει ο καθένας να σέβεται, να γνωρίζει τον άλλον και να καταλάβουμε ότι ο αλληλοαποκλεισμός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβραδύνει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένταξης. Για το περιβάλλον. Νομίζω ότι αυξάνει όλο και περισσότερο σε σημασία. Θέλουμε μια υφόρο ανάπτυξη, αλλά να έρθουμε και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις διαφορετικές ιδέες και τα σημαντικά προγράμματα που έχουμε στο μέλλον, όλα αυτά θα εξετάζονται πρώτα απ' όλα από ε, πλευράς περιβαλλοντικού αντικτύπου. Γιατί θέλουμε και στην να συναπούμε και να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Και για να αναπτύξει κάποιος τον τουρισμό χρειάζεται ένα περιβάλλον το οποίο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να φροντίζουμε τα έργα να ε, ε, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να μην το προσβάλλουν. Για τις καθυστερήσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αν φταίει κάποιο κόμμα, κάποια πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω εδώ να ζητάω, να ψάχνω εχθρούς. Όπως είπε ο κύριος Βένσον όμως, είναι γεγονός αυτό. Πριν από μερικές δεκαετίες και μόλις πριν από 20 χρόνια η Αλβανία ήταν η Βόρεια Κορέα της Ευρώπης. Η πιο απομονωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μέσα σε δύο και μόνο δεκαετίες είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και έχουν προχωρήσει οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε ένα τέτοιο στάδιο που σίγουρα θα ενταχθεί η Αλβανία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι χρονικό τώρα βεβαίως και αυτό θα εξαρτηθεί από τις εσωτερικές μας μεταρρυθμίσεις αλλά και από τη βούληση και τα βήματα που θα κάνει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μελλοντική της διεύρυνση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε ότι θα πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει ε, στη επιτάχυση της διαδικασίας αυτής. Και το θέλει και το Κοινοβούλιο και η αντιπολίτευσή μας. Γιατί και το Σοσιαλιστικό Κόμμα συνεισέφερε τα μάλα στο παρελθόν για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Σχετικά με την ερώτηση τώρα, εάν οι ηγέτες του Δημοκρατικού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουν συναντηθεί, νομίζω ναι. Στο παρελθόν επανειλημμένος. και με πλήρη συνένεση έγινε αλλαγή στον εκλογικό νόμο, κάποια συνταγματική ενθεώρηση και θα ήταν πολύ χρήσιμο επίσης και θετικό να ε, ξαναδούμε τέτοια συνεργασία για το συμφέρον της χώρας και της ευρωπαϊκής ατζέντα της Αλβανίας. Σε σχέση με το ε, εμπόριο ανθρώπων είναι βεβαίω ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά μειώνεται όλο και περισσότερο το πρόβλημα γιατί η ε, κυβέρνησή μας εμφανίζει μια ισχυρή βούληση και τώρα έχουμε άριστη συνεργασία με ε, τις γειτονικές μας χώρες και η Αλβανία δεν είναι πλέον χώρα ε, διέλευσης για το τράφικινγκ. Συνεργαζόμαστε περιφερειακά για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα δουλείας και γι' αυτό αναλαμβάνουμε και την πρωτοβουλία προσεχώς να διοργανώσουμε οργάνωση, ε, ε, διάσκεψη συγγνώμη, για την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνάντηση για να μάθουμε όλα τα θετικά επιτεύγματα της χώρας σας, αλλά και τα κολλήματα για την προσχώρηση της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε, θα αξιοποιήσετε όλες τις αναφορές που έγιναν εδώ για να προχωρήσετε στην προσέγγιση της χώρας σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 10.30 συνεχίζουμε για να ψηφίσουμε. prezli risk uh, Καθίστε, παρακαλώ πολύ, θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Καθίστε, παρακαλώ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ να βάλετε ήδη την καρτούλα σας στο μηχάνημα για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί καλά. Ξεκινάμε με τα δοκιμαστικά. Πατήστε ένα κουμπάκι να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Είμαστε 34 παρόντες. 34 φαίνεται. Beh, ci sono alcuni ε, φαίνεται ότι είναι μερικοί συνάδελφοι που δεν κάνουν τη δοκιμή. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε το τεστ να δούμε αν δουλεύει το μηχάνημα. Βάζοντας την καρτούλα σας στο σχετικό μηχανάκι και πατώντας το κουμπί. Όποιο κουμπί θέλετε. Ωραία. Τελειώσα. 45 παρόντες. Έχουμε και η δοκιμή ήταν πολύ μικρότερη, με μικρότερο αριθμό. Ψηφίζουμε την έκθεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράγραφος 1, τροπολογία 27, δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 28 του συγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει η προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε την 29, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Δεν κατάλαβα. Δεν είδα πολλά χέρια στον αέρα. Ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 30 αρχίζει η ψηφοφορία. 59 κάρτες είναι στα μηχανήματα, 49 ψήφισαν. 36 υπέρ, 12 κατά. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά εγκρίνεται. 34 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 34 και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. 34 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά μου φαίνεται να απορρίφθηκε 35 λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 22-34 απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά απορρίπτεται 44 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβασμός 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 50 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται 51 υπέρ κατά απορρίπτεται 52 έχει καταπέσει όχι δεν έχει καταπέσει ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται 53 του συγητή Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 52 αρχίζει ψηφοφορία. «57 ψηφίσαντες, 30 κατά, 25 υπέρ. Απορρίπτεται 53 του εισηγητή υπέρ. Κατά εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έχει καταπέσει 56. Διότι δεν πέρασε 43. 57 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8, συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά εγκρίνεται 75 υπέρ Εβδομήντα πέντε λοιπόν έλεγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα εφτά υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 79 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 80 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 81 έχει αποσυρθεί, 82 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ κατά, αποχές, 84 έχει καταπέσει, 85 υπέρ, 86 έχει καταπέσει, 88-89 είναι ίδιες. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 έχει καταπέσει 91 υπέρ κατά εγκρίνεται 92 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 έχει καταπέσει Προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά απορρίπτεται 99 υπέρ κατά εγκρίνεται 100 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται <coughs> Νέο συμβιβασμό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 102 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά εγκρίνεται 106 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβασμός 9 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στην 112 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται 113 υπέρ κατά εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά απορρίπτεται 116 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 117 υπέρ κατά εγκρίνεται Εθιμώντας α, 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 24 του εισηγητή υπέρ. Η εισηγήτρια θέλει το λόγο πριν από την έγκριση της τροπολογίας 24. Έχετε το λόγο κυρία Χάουταλα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια προφορική τροπολογία μετά από συζήτηση που έγινε με συναδέλφους να προσθέσουμε το ότι έχουμε εδώ πέρα εντοπίσει πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μπει η φράση «on the position of extensive fines». Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, ψηφίζουμε την τροπολογία ούτως διατυπωμένη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τίτλος 1. Είναι γλωσσική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέσσερα, Υπέρ. πέντε, Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Έξι, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, είναι η τελική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. 64 παρόν, 65 παρόντες, 63 ψηφίσαντες πέρας ψηφοφορίας. 59 υπέρ, ένας ε, κατά και τρεις αποχές. Ε, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εγκρίνεται η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Είναι λίγο μπερδεμένα εδώ τα πράγματα. Ελπίζω να μην ε, κάνουμε πολλές ε, ζημιές. Λοιπόν, έχουμε βέβαια πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σα. Παράγραφο 1. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Εγώ θα έλεγα απορρίφθηκε. Έχει καταπέσει 91. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, έχει καταπέσει, έχει καταπέσει, γιατί ψηφίσαμε το συμβιβασμό, σωστά. 102 λοιπόν, υπέρ, κατά, εδώ δεν κατάλαβα καλά. Λυπούμε, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 102. Αρχής ψηφοφορία. 65 votanti, 64 voti espressi. 64, 65 έχουν ψηφίσει. 31 υπέρ και 33 κατά έχει απορριφθεί. 103 εγκρίθηκε ο συμβιβασμός 4. 104 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 107 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 108 που είναι συμβατή με την 5 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 111. Καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 28, 112 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Αποσύρεται 113, περνάμε στην 114 του συγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 122 του συγητή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 128 συνάδει με την 6 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 130 παρά με συμβαστική 27 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Γλωσσική αλλαγή στην 136 ψηφίσουμε 137 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 του συγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. ηλεκτρονικός έλεγχος για την 140 άρχιτη ψηφοφορία. Εξήντα 64 ψηφίσαντες, 14 υπέρ, 46 κατά, απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 142 και 143 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 144 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 145 αποσύρεται. 146 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα της 146 άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, έλεγχος. ...62 ψηφίσαντες, 28 υπέρ, 32 κατά. Δύο εποχές. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Αποσύρεται η τροπολογία 148 και προχωράμε με τις 149 και 150 υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Συμβαστική προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 151 για την απλώς γλωσσική αλλαγή 152 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 156 και 157 υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 169 καταπίπτει γιατί ψηφίσαμε τη συμβαστική 10, 170 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 175 καταπίπτει, όπως και 176 και 177. Περνάμε λοιπόν στην συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 203 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 214 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 225 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 225, άρχιτη ψηφοφορία. «66 ψηφίσαντες, 31 υπέρ, 35 κατά, απορρίπτεται». 226 με την προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 22 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει και περνάμε στην συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 38 συμβατή, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 39 με την προφορική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Υπέρ εγώ νόμιζα ότι είδα, αλλά δεν σήκωσαν όλοι τα χέρια τους ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 45 άρχιτη ψηφοφορία. «62 ψηφίσαντες, 42 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, δεν μπορώ να πω, γιατί 47 α, θα είναι καλύτερο να ελέγξουμε, πιστεύω, γιατί δεν α, σηκώστε τα χέρια σας. Λοιπόν, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 47. 62 ψηφίσαντες. Ναι, ναι, βλέπω ότι είναι μεγάλη η πλειοψηφία, 56 προς 6. Λοιπόν, θα αλλάξω γυαλιά, λέει ο πρόεδρος. 48, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 49, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 50, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αποσύρεται 52, περνάμε στην 53 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά, εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 66 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 67 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 68 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 69 υπέρ κατά απορρίπτεται. Αποσύρε... Αποσύρθηκε η 70, 71 υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έχει καταπέσει. 74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. 75 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 53 υπέρ, εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά εγκρίνεται 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 3 αποσύρθηκε 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται Λοιπόν, έχουμε ψηφοφορίες από την Επιτροπή Διεθνού Συμπορίου. Έχουν καλυφθεί οι πρώτες, οπότε ψηφίζουμε την 7, υπέρ. Κατά εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά εγκρίνεται 10 υπέρ, κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται η κυρία Φλότρα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε θα έλεγα θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε στην παράγραφο 13 που αφορά στην γεωργία της κυρίας Δεσαρνές είναι αλήθεια ότι έχουμε και την 11 για τη Γεωργία, αλλά εδώ προτείνεται κάτι το οποίο δεν είναι ασύμβατο, προτείνω να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Πεγιόν τι λέει. Θεωρούσαμε ότι καλυπτόταν, υπάρχουν μερικές βέβαια ε, διαφορές, είμαι υπέρ, υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν την ίντα 13, υπέρ. υπέρ κατά εγκρίνεται. Είναι το 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ήτρε. Ήτρε 1 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Ήτρε 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ήτρε 9 υπέρ κατά εγκρίνεται, ήτρε 10 υπέρ, κατά εγκρίνεται, ήτρε 13 υπέρ, κατά εγκρίνεται, ήτρε 14 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τσεκ ε, για την ήτρε 13. Ε, όλα είναι δυνατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία ήτρε 13. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. Ήτρα 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρα 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρα 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία αρχίζει ψηφοφορία. Εξήντα τέσσερις ψήφισαν. Εξήντα πέντε, μάλλον, εξήντα πέντε. 58 λοιπόν υπέρ, 6 κατά εγκρίνεται ε, η έκθεση. Συγχαρητήρια. Πέρας ψηφοφορίας, ξαναπάρτε τις κάρτες σας. 11.30 με την ακρόαση του Επιτρόπου Φιούλε. Ο κύριος Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, και στην έκθεση αυτή πάλι γράψαμε ε, σημαντική αύξηση των πόρων στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και αν συνεχίσουμε έτσι φοβάμαι, σε όλες τις εκθέσεις ανεβάζουμε τα λεφτά. Να το σκεφτούμε. Ε, πού θα έχουμε βρεθεί όταν φτάσουμε πραγματικά στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και αν έχουμε βάλει παντού παραπάνω διακυβεύεται πολύ η αξιοπιστία μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια φόρμουλα πώς θα το αντιμετωπίσουμε για να παραμείνουμε συνεπείς και να μας παίρνουν και σοβαρά. E- Ευχαριστώ τον κύριο Μπροκ. Συνεχίζουμε στις 11.30 με τον Επίτροπο Φίλε.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 Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στη ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον φίλο και συνεργάτη τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης, Στέφαν Φούλε, ο οποίος πρόσφατα πήγε στον Νότιο Κάυκασο στις αρχές Απριλίου και την προηγούμενη εβδομάδα πήγε στην Ουκρανία. Εξ όλων πρέπει να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευαισθησία που δείχνει απέναντι στη δική μας Επιτροπή και γενικότερα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εμείς εκπροσωπούμε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι έρχεται εδώ πέρα για να μας μιλήσει άμεσα για τις εντυπώσεις που είχε από την επίσκεψή του αυτή και για να μας μιλήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ε, χώρες αυτές, ιδίως σε σχέση και όλες με τις πρόσφατες εκλογές στην Ουκρανία. και ξέρετε ότι αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την χώρα αυτή και με τις υπόλοιπες χώρες του Νότιου Καυκάσου. Έχουμε και το ζήτημα της διαπραγμάτευσης ε, των ε, συμφωνιών σύνδεσης με την ε, Ουκρανία και την απαρχή των διαπραγματεύσεων αυτών για τον Νότιο Κάυκασο. Το απόγευμα θα έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με αυτά τα σχέδια διαπραγματευτικών οδηγιών για τις συμφωνίες ε, σύνδεσης. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό. Έχουμε και την πρόσφατη έκθεση από τον συνάδελφο Κύριλοφ, την οποία εγκρίναμε στην Επιτροπή μας. Δεν θα ήθελα να αφαιρέσω άλλο χρόνο από τον Επίτροπο και από τους συναδέλφους, επομένως ευθύς αμέσως του δίνω το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που είπατε ότι δεν πρόκειται για μία απομονωμένη περίπτωση ad hoc εμφάνισή μου εδώ είναι μέρος της αρχικής συμφωνίας που είχαμε κάνει. Από τότε ανέλαβα τις αρμοδιότητές μου να έχουμε δηλαδή μια διαδραστική σχέση συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματική τιμή για μένα να μοιραστώ μαζί σα ε, τι εντυπωσει μου από την επίσκεψη που είχα στι τρει ε, χώρε του Νοτιού Καυκάσου καθώ επίση και στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με τον Νότιο Κάυκασο. Θα ήθελα να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων μετά την δική σας ε, έγκριση στην έκθεση που έχετε για τον Νότιο Κάυκασο, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι πολλές από τις συστάσεις, της, ε, πολλές από τις συστάσεις αυτής θα συμφωνήσουν με αυτά που θα πω σήμερα. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρώπη άκουσα από το ταξίδι που έκανα στην Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν. Οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι κυβερνήσεις αλλά και η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών όλοι επιβεβαίωσαν ότι θέλουν μια στενότερη, βαθύτερη και πιο πλήρη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα λοιπόν προς τους συνομιλητές μου στην Γερεβάν, την Πακού και την Τυφλίδα ήταν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιταχύνει και να ενισχύσει, να ενισχύσει με συγχωρείτε, τους τομείς εκείνους όπου μπορούμε να έχουμε μια πιο ενισχυμένη συνεργασία και σχέση με τους λαούς του Νοτίου Καυκάσου. Στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης που ξεκίνησε πέρυσι στην Πράγα, είμαι πεπισμένος ότι το σχέδιο αυτό συνεργασίας μπορεί να επιτύχει σε πάρα πολλά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις που έχουμε με τους εταίρους μας προς Ανατολάς. Με την Ουκρανία, στην οποία θα αναφερθώ λίγο αργότερα, έχουμε ήδη διαπραγματευτεί μια συμφωνία σύνδεσης πριν από δύο περίπου χρόνια και έχουμε και διαπραγματεύσεις με την ε, Μολδαβία οι οποίες ε, ξεκίνησαν σε αρχές του 2010 και συνεχίζονται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Χαίρομαι που σας λέω σήμερα ότι ε, οι οδηγίες διαπραγμάτευσης με, για τις συμφωνίες σύνδεσης με τις ε, χώρες του Νοτιού Καυκάσου θα παρουσιαστούν το, στις 10 Μαΐου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προετοιμαστεί για την επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι συμφωνίες αυτές θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ε, έντονη πολιτική εταιρική σχέση με τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, που η οποία θα βασίζεται σε κοινέ αρχές. Και αναγνωρίζω βέβαια τον πολύ σημαντικό ρόλο που διδραματίζει η δική σας Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει βαθείς και πλήρης σχέσεις ελευθέρων συναλλαγών με τις χώρες αυτές. Και εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, ιδίως για τις χώρες εκείνες του Νοτίου Καυκάσου που πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρόκειται για συμφωνίες οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως ονομάζω, που θα δώσουν πρόσβαση στις χώρες αυτές στην πολύ μεγάλη αγορά καταναλωτών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται όμως απλώς για εμπορικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές θα οδηγήσουν σε μία ευθυγράμμιση όσον αφορά το κοινοτικό κεκτημένο για το εμπόριο και την ιστορική αγορά. Όσον αφορά τώρα τις θεωρήσεις και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών. Και εδώ η εταίροι μας στον Νότιο Κάφκασο ζητάνε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιώθουν πλέον την πίεση των πολιτών τους που θεωρούν ότι οι διαδικασίες είναι πολύ πολύπλοκες και μακροχρόνιες. Η διευκόλυνση λοιπόν του καθεστώτος θεωρήσεων και οι α, συμφωνίες επανεισδοχής έχουν ήδη κλείσει με επιτυχία για την Γεωργία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι Γεωργιανοί θα έχουν χαμηλότερα τέλη και πιο εύκολους κανόνες χορήγησης θεωρήσεων. θα θέλαμε ανάλογες ε, διαπραγματεύσεις και με τις υπόλοιπε χώρες του Νοτιού Καυκάσου. Αυτό επιθυμούν τουλάχιστον οι πολίτες από την Αρμενία και το Ζερβαϊτζάν. Σίγουρα οι ε, απαιτήσει είναι πολύ σημαντικές από πλευράς χωρών Νοτιού Καυκάσου, αλλά εξίσου σημαντικές ε, είναι οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε να υπάρχουν οι απαραίτητες νομοθεσίες, καθώς επίσης και απαραίτητη διοικητική υποδομή, προκειμένου να μπορούν οι χώρες αυτές να οδηγηθούν σε απτά αποτελέσματα στα πλαίσια των συμφωνιών που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τους ηγέτες τη Αρμενίας, του Αζερβαϊτζάν και της Γεωργίας, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε είναι ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες μεταρρύθμισης και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και ότι βέβαια γι' αυτά ευθύνονται οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί στις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τεχνική και χρηματοοικονομική αρρωγή προς τις χώρες αυτές προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, ιδίως ε, μέσω των ε, νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων ε, οικοδόμησης θεσμών που έχουμε διαπραγματευτεί με τις χώρες αυτές. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να σας πω ότι Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές και προσπαθούμε να πετύχουμε τις χώρες αυτές μια βαθύτερη και στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αρμενία ζήτησα από όλου του πολιτικού ηγέτε να γίνουν οι απαραίτητε πολιτικέ μεταρρυθμίσει προκειμένου να αλλάξουν τα στάνταρ για τι εκλογέ και προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν κάποια από τα πολιτικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν μετά τι προεδρικέ εκλογέ του Μαρτίου του 2008, προκειμένου να υπάρχει εθνική συμφιλίωση στη χώρα και προκειμένου να μπορεί η κοινωνία να λειτουργήσει πλήρως. Με άλλα λόγια, ζητήσαμε, συζητήσαμε πολύ το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Γεωργία και ιδιαίτερα τις επερχόμενες τοπικές εκλογές τον Μάιο, είχα τη δυνατότητα να ακούσω και τους κυβερνητικούς εκπροσώπους αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και στις δύο πλευρές είπα ότι θα πρέπει να προσχωρήσουν στις διεθνείς προδιαγραφές για τη διεξαγωγή των εκλογών, ότι πρέπει να υπάρχει πολιτικός πλουραλισμός και ότι θέλουμε μια ζωηρή κοινωνία των πολιτών η οποία να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά και ότι αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εδραιωθεί η δημοκρατία. Με άλλα λόγια, πρέπει να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, το ότι δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δημοκρατικές δυνάμεις αφενών, αφενός και τις κοινωνίες των πολιτών αφετέρου, των υπόλοιπων δυνάμεων του πλουραλισμού. Για το Αζερβαϊζάν ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένας διάλογος πλέον ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας αυτής, προκειμένου να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και σε άλλους τομείς πέρα από τον τομέα της ενέργειας. Συμφωνήσαμε ότι ε, η... Το βασικό, ο βασικός τομέας συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν είναι όντως η ενέργεια. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η οικονομία της χώρας και να ενισχυθούν περισσότερο οι περιφέρειες, οι επαρχίες της χώρας. Ζητήσαμε επίσης περαιτέρω προσπάθειες εκδημοκρατισμού και μεγαλύτερο συμβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες αυτό που συζητήσαμε τόσο με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών, συγγνώμη, τον Πρωθυπουργό, ήταν να καταφέρει να δεσμευτεί στους τομείς αυτούς επίσημα πλέον το Αζερβαϊζάν. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντα στο Νότιο Κάφκασο, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια συνεχόμενη πολιτική ένταση στην περιοχή και συνειδητοποίησα επίση πολύ οδυνηρέ επιπτώσει των τοπικών διενέξεων στου ε, πληθυσμού εκεί. Στο Αζερβαϊτζάν και στη Γεωργία μίλησα με εκπροσώπου εκτοπισμένων πληθυσμών και συνειδητοποίησα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνει η Επιτροπή Επιτήρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από την Τυφλίδα. Οι προσωπικές αυτές ιστορίες προσωπικής τραγωδίας ουσιαστικά με βοήθησαν να καταλάβω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του Νότιου Καυκάσου. Οι διενέξεις αυτές έχουν επισκιάσει πλέον τον Νότιο Καύκασο και τη ζωή των πολιτών για πάρα, πολλά, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και επαναλαμβάνω την βασική επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει πλέον ειρήνη, σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Όσον αφορά τώρα την ομαλοποίηση των σχέσεων Αρμενίας-Τουρκίας, και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Και ότι καταγράφω τις τελευταίες εξελίξεις προηγούμενης εβδομάδος, Λέω ότι η Αρμενία παραμένει δεσμευμένη να συνεχιστεί η διαδικασία όσον αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει την υποστήριξή της στις ειρηνευτικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη. Όσον αφορά τη Γεωργία, είναι σαφές ότι οι συζητήσεις της Γενέβης είναι πολύ σημαντικές προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρεθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι συζητήσεων και προκειμένου να καταφέρουν να προλάβουν νέες κρίσεις στο μέλλον. Είναι σημαντικό να δεσμευθεί η Γεωργία όσον αφορά την πρωτοβουλία συνεργασία την οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα την Ουκρανία, πήγα στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα πολλέ χρήσιμε επικοδομητικέ συναντήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, μέλη τη Αντιπολίτευση και εκπροσώπου από επιχειρήσει και την κοινωνία των πολιτών. η επίσκεψη ερχόταν σε συνέχεια επίσκεψη της ΥΠΑ της εκπροσώπου και δικής μου α, επίσκεψης, καθώς επίσης και μετά από την επίσκεψη του κυρίου Γιαννούκοβιτς στην Βρυξέλλες την 1η Μαρτίου. Θέλησα να μιλήσω με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και με τους επικεφαλείς από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και με τον Μπόρι Σταρασούκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή η επίσκεψη αυτή, γιατί ουσιαστικά συνέπεσε με τις προτιμασίες της κυβέρνησης προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα μεταρρύθμισης, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και ήρθε την κατάλληλη στιγμή επειδή υπήρξε μία ανακοίνωση όσον αφορά το φυσικό αέριο αλλά και την παρουσία του ρωσικού στόλου παρουσίασα στην ε, ρωσική πλευρά τις βασικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η Ουκρανία και ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά κίνητρα τα οποία θέλει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατάλογος αυτός καλύπτει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, μακροοικονομική σταθερότητα, ένα κατάλληλο περιβάλλον για το εμπόριο και την οικονομία, κινητικότητα και καλύψαμε και το ζήτημα της ενέργειας. Με πολλές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας συνεργάστηκα και βασίστηκα επίσης και συζητήσεις που έχουν γίνει στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Θα σας δώσω λοιπόν το έγγραφο αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχετε κι εσείς τον πίνακα αυτό και να δείτε πώς ουσιαστικά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε τους δύο καταλόγους. Έναν κατάλογο με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, απαιτούμενες από την Ουκρανία μεταρρυθμίσεις, και έναν κατάλογο με τα κίνητρα τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. και η ε, επίσκεψή μου επί τόπου πραγματικά με βοήθησε να καταλάβω πώς ε, η κυβέρνηση στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια προχωρά με τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Ο πίνακας αυτός λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα αποτελέσει ένα εύχριστο εργαλείο προκειμένου να κατευθυνθούν καλύτερα τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της ε, κυβέρνησης και να διατηρηθεί ένας καλός ρυθμός στα προγράμματα μεταρρύθμισης θα βοηθηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η Ουκρανία περισσότερο στο δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και θα βασιστούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στις προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί και στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης. Θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καθοδηγήσουμε πολιτικά τις μεταρρυθμίσεις στην ε, χώρα. Δεν αποτελεί ο πίνακας αυτός που σας δίνω επίσημο τμήμα της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης και των σχετικών συζητήσεων. Πρόκειται για ένα κοινό εργαλείο που έχουμε, Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή αφενός και οι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου είναι συμβατές. Ότι πρόκειται για δύο συμβατές διαδικασίες, όχι μόνο σε αρχικό στάδιο, σε θεωρητικό στάδιο, αλλά και στο στάδιο της εφαρμογής. Όσον αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης, εκφράστηκε η πρόθεση να υπογραφεί η συμφωνία αυτή το 2010. Σας υπενθυμίζω ότι σκεφτόμαστε αρχικά το 2011 ως προθεσμία και ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς το είπαν αυτό την 1η Μαρτίου. Εγώ εξήγησα ότι χρειαζόταν ακόμα περισσότερη δουλειά, ιδίω όσον αφορά τη δημιουργία ελεύθερη όνη συναλλαγών από ουκρανική πλευρά, αλλά από την άλλη τόνισα ότι θέλουμε κι εμεί να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει σύνδεση στο συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά τώρα το διάλογο για τι θεωρήσει, εξήγησα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια προσέγγιση οδικού χάρτη για τις θεωρήσεις, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες βελτιώσεις από ουκρανικής πλευράς. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης γίναν κάποιες αρχικές συζητήσεις με τους ε, υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν. Περιμένουμε όμως μεγαλύτερη πρόοδο ακόμα από την Ουκρανία και περιμένουμε να δούμε πιο απτά αποτελέσματα στη σύνοδο που θα γίνει το φθινόπωρο. Είπα επίσης ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη στρατηγική, μια καλύτερη στρατηγική ολοκλήρωσης και ενσωμάτωση όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και όσον αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις της ε, χώρας. Ο Μπόρις Τάρατσουκ αλλά και ε, η πρώην Πρωθυπουργός Τιμοσέγκο συμφώνησαν με αυτό. Έδωσα τον πίνακα τον οποίο σας έδωσα και στους ε, ηγέτες αντιπολίτευσης και τους εξήγησα ότι θα πρέπει στα πλαίσια του κοινοβουλίου τους να συνεργάζονται περισσότερο προκειμένου να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ενημερώθηκα επίσης για τη νέα συμφωνία φυσικού αερίου με τη Ρωσία και επίσης ενημερώθηκα για την ε, παρατεταμένη παρουσία του ρωσικού στόλου στην Κρυμαία. Ξέρετε ότι τα ζητήματα αυτά είναι αρκετά διαφιλονικούμενα και υπάρχει έντονη αντιπαράθεση σε εσωτερικό επίπεδο στη χώρα. Καταλαβαίνω τώρα γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε επανεδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας για το Φυσικό Αέριο. Μετά τις, τα γεγονότα του 2009 έπρεπε σαφώς να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα παροχής ενέργειας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εγκρίνει προπολογισμό για το 2010 και να ξεκινήσει πλέον συνομιλίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάσει νέων δεδομένων. Παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση επέκρινε την παρατεταμένη παρουσία του ρωσικού στόλου στην Κρυμαία και θεώρησε ότι πρόκειται για μια παραχώρηση που γίνεται ακόμα και σε θέματα κυριαρχίας. Όσον αφορά το φυσικό αέριο θα εξεταστεί η συμφωνία περισσότερο και αυτό τόνισα και εγώ στο Κίεβο. Θα εξεταστεί από, την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί σαφώς η τροφοδοσία με σε φυσικό αέριο, ότι θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη προβλεψιμότητα και διαφάνεια και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο εξυγχρονισμός του συστήματος παροχής φυσικού αερίου. Όσον αφορά τώρα την κυριαρχική διάσταση της συμφωνίας αυτής για την Ουκρανία, είπα ότι θα πρέπει η διαπραγμάτευση αυτή να γίνει στα, πλαίσια του, στα συνταγματικά πλαίσια της χώρας. Τι αποκόμισα ε, από την επίσκεψη αυτή, ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για τη νέα ε, κυβέρνηση. Έχει στείλει σαφή μηνύματα ότι είναι προσιλωμένη στην ευρωπαϊκή ολοκληρωσία και στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Θα μάθουμε πολύ περισσότερο για αυτά τα θέματα μόλις ε, τον Ιούνιο καταθέσει η νέα κυβέρνηση το μεταρρυθμικό πρόγραμμα. Η ε, μήτρα για τις μεταρρυθμίσεις όπως και άλλα ε, θέματα, η διαδικασία και τα θέματα για τη σύνδεση θα μας επιτρέψουν να δούμε κατά πόσο οι υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται και από δράσεις και από λόγια και από έργα, συγγνώμη. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητε μου του επόμενου μήνες. Ε, στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να ε, συνεργαστεί με την Ουκρανία εάν και ε, όταν εφαρμόσει εκείνη τη μεταρρύθμιση. Σας έχω δώσει παραδείγματα πιθανές αποκρίσεις ποιες ε, μπορεί να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θετικά μηνύματα. Αυτό αρχίζει ε, από ε, οικονομική βοήθεια, οικονομική βοήθεια μέχρι πρόοδο στην κινητικότητα και μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε όχι μόνο με την κυβέρνηση, αλλά και με άλλους βασικούς φορείς της χώρας και μεταξύ αυτών το Κοινοβούλιο. Ε, με μέλη της αντιπολίτευσης, με ε, εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι μια διαδικασία συμπερίληψης. Με ενθάρρυνε η προσήλωση και της αντιπολίτευσης στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν ε, πιο κοντά την Ουκρανία στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συνεχίζουμε λοιπόν τις προσπαθίες μας στο Νότιο Κάφκασο και στην Ουκρανία και με τη γειτονία και έτσι πιστεύω ε, ότι θα μπορέσει και το Κοινοβούλιο σας, η Επιτροπή σας και η Κοινοβουλευτική Συνεργασία και οι διάφορες επιτροπές να παίξουν ένα πολύ ε, πολύτιμο ρόλο. Και θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε όπως είχαμε και σήμερα. Σύμφωνα με την πρακτική ε, προηγουμένων ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί ε, τις ε, εξελίξεις στις γειτονικέ χώρες μέσω των ετησίων εκθέσεων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Οι φετινές εκθέσεις γειτονίας θα είναι ένα μείγμα επένων αλλά και υποδείξεων όταν χρειάζεται και περαιτέρω πρόοδοι για προγράμματα δράσης προσβλέπω να επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 του μήνους Μαΐου, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση των εκθέσεων της γειτονία για να συζητήσουμε τα μελλοντικά μας σχέδια μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ήταν μια συνάντηση, τουλάχιστον στο εισαγωγικό της μέρος, πολύ ενδιαφέρουσα. Να δούμε τώρα στη συνέχεια αν η συζήτηση θα είναι και αυτή στο ύψος ε, των ε, ευθυνών που μας εμπίπτουν. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για τον Νότιο Κάφκασο, τον κύριο Κυριλόφ. Τρία λεφτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, φίλε, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις ε, πρωτοβουλίες που αναλάβατε τόσο νωρίς και τις επισκέψεις. Ε, ως εισηγητής για τον Νότιο Κάφκασο πρέπει να σας πω ότι έχω ήδη πληροφόρηση ε, το εκτίμησαν πολύ το γεγονός ότι πήγατε τόσο γρήγορα εκεί και αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και για την επίλυση θεμάτων ασφαλείας ε, και για το ενδιαφέρον για τη συνεργασία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γνωρίζετε ότι εδώ και καιρό δεν έχουμε ισχυρή παρουσία εκεί. και τα μηνύματα είναι εκείνα που θα μας ε, βοηθήσουν να ενεργοποιήσουμε την πολιτική μας και πραγματικά μας χρειάζονται πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή σας στις τρεις χώρες του Νοτιού Καυκάσου, αυτές συνδέονται με μία υπόσχεση ότι ενεργούς ε, ανάπτυξης ε, των σχέσεών μας με τις χώρες αυτές και τη σταθεροποίηση. Βεβαίως είναι και θέμα δημοκρατισμού. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πολύ στενές, σοβαρές ε, και επιμερούσες σχέσεις με τις χώρες αυτές. Είμαι βέβαιος ότι θα διαπιστώσατε ότι κάθε χώρα ε, χρειάζεται βέβαια ξεχωριστή μεταχείριση, αλλά εμείς προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε και τις τρεις από κοινού και να ενθαρρύνουμε και ε, διαπεριφερειακή μεταξύ τους συνεργασία για να συνεισφέρουμε για τη σταθερότητα της περιοχής. Τι με ενισχύει τώρα εμένα και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου. Οι δύο σειράξεις και οι ε, Ρωσογεωργιανοί που περιμέναμε μέχρι να ξεσπάσει και τώρα είμαστε και παρόντες βέβαια, αλλά και η άλλη σύραξη, η σύγκρουση που δεν έχουμε σαφή θέση για το ορεινό Καραμπάχ. Λοιπόν και, και οι δύο περιπτώσεις χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή και την προσοχή μας και την συμμετοχή μας κατά κάποιο τρόπο εκεί. Εδώ στην Επιτροπή μας συζητήσαμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε με εντολή για την πρόοδο των διαγραμματεύσεων ε, γιατί η συνδίκτηση Λισαβόνας δεν μας επιτρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε απλοί παρατηρητές. Τι έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, ύψη σημασία. Αυτά οι δύο σύγκρουσει επισκιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Έχουν πολύ μακριά σκιά. Και όχι μόνο τα οικονομικά θέματα, αλλά και τα δημοκρατικά θέματα και τη δημοκρατική πρόοδο. Και είναι ε, ζωτική σημασία. Τελειώνω λοιπόν, κύριε Φίλερο, λέγοντα το εξή. Σε σχέση με αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το συζητήσετε με τη Λέδη Άστον. Πρέπει να πάει εκεί γρήγορα η Λέδη Άστον και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Διότι να κάνουμε απλώς δηλώσεις για τις αρμενοτουρκικές σχέσεις δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυριλόφ. Ο συνάδελφος Κόβατσεφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση όσον αφορά την επίσκεψή σα στην Ουκρανία και τον Νότιο Κάυκασο. Πολύ σημαντική συνεργασία αυτή που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής μας. Ένα ζήτημα όσον αφορά την Αρμενία και τις σχέσεις Αρμενίας και Τουρκίας τόσο για το ζήτημα των συνόρων, καθώς επίσης και για τα, την 25η επέριουσαστικά της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία θέλουν να ολοκληρώσουν συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε εμείς να εμπλακούμε πιο ενεργά με τρόπο θετικό ώστε να επιλύσουμε τις διενέξεις αυτές ανάμεσα στην Αρμενία και το Ζερμπαϊτζάν και την Αρμενία και την Τουρκία. Και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την Ουκρανία, καθότι εξ ονόματος του ΕΛΚ ασχολούμαι με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Είπατε σε επίσκεψη πανεπιστήμιο της χώρας ότι ένα 90% της εξωτερικής πολιτικής της χώρας συνάδει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι όμως πολιτικοί αναλυτές λένε ότι βλέπουν ότι η εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας αρχίζει να στρέφεται περισσότερο προς την Ρωσία. Τι πιστεύετε εσείς, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο μέλλον, αυτό το 90% θα αυξηθεί, ή θα μειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόβατσεφ. Κύριο Στάλερ για δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα... Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δράση σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ευρωαλληλική περιοχή της Υπήρου μας. Πριν από ένα μήνα είχαμε συναντηθεί στην Τυφλίζα μαζί, 12η ε, κατά σειρά ήταν η συνεδρίαση που είχαμε. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, κάναμε κάποιες συστάσεις εκεί Το Δεκέμβριο είχαμε αντίστοιχη συνάντηση στο Αζερβαϊτζάν και προσεχώς ε, ε, πήκεται η Αρμενία. Και οι τρεις αυτές χώρες ενδιαφέρονται πολύ να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά αυτό για τη σταθεροποίηση της περιοχής ολόκληρης. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Σε σχέση ακριβώς με τις τελευταίες συγκρούσεις εκεί στην περιοχή. Η συγκεκριμένη σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας πώς αξιολογείται τη σημερινή κατάσταση. Τη συνομιλία της Γενέβης και βλέπετε να έχει κανένα πιο ενεργό ρόλο να διδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειες να στεφθούν με επιτυχία αυτές οι συνομιλίες. θα πρέπει να επενέσουμε την ε, Επιτροπή την αποστολή παρακολούθησης και παρατήρησης που έχουμε εκεί. Γιατί είναι πολύτιμη συνεισφορά για την παρακολούθηση των προβλημάτων και των εξελίξεων. Βλέπετε καμία δυνατότητα συμφωνίας έτσι ώστε ε, να μπορεί να περνάει και τα σύνορα. Για δύο λεπτά ο κύριος σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα ερώτημα σχετικά με την επίσκεψη στην Ουκρανία. Η Ουκρανία στο παρελθόν κοιτούσε δυτικά, τώρα κοιτάει περισσότερο ανατολικά Γίνανε κάποιες αναφορές όσον αφορά την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ που δεν την προωθεί πλέον η Ουκρανία. Πρέπει όμως να ληφθεί περισσότερο υπόψη το θέμα της ασφάλειας. Η παρουσία για παράδειγμα του ρωσικού στόλου στην Κρυμαία. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα της ασφάλειας όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Ξέρουμε ότι ανατολικά και δυτικά της Ουκρανίας η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Έχετε εσείς την εντύπωση ότι η Ουκρανία είναι ουσιαστικά διχασμένη όσον αφορά το μέλλον της ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Βαμπάλεν, ο κύριος Σούλτς για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, φίλε, αναφερθήκατε σύντομα μόνο στη σημερινή σύραξη που ε, πλήττει περισσότερο ακόμα μια διαιρεμένη χώρα. Η ε, παράταση της στρατιωτικής ε, ε, συμφωνίας για 25 ακόμα χρόνια με τη Ρωσία, για το στρατό, το στόλο μάλλον το ρωσικό που σταθμεύει στην Κρυμαία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πάει πολύ μακριά τώρα η ένταξη ενδεχόμενη της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρική είναι για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις επισκέψεις σας στις τέσσερις αυτές χώρες που αποτελούν τμήμα της πολιτικής γειτονίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ουκρανία θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σας αξιολόγηση όσον αφορά την απόφαση του Κοινοβουλίου να παρατείνουν την δυνατότητα παραμονής του ρωσικού στόλου στην Κρυμαία για πέντε επιπλέον χρόνια μετά το 2017. Είδαμε τι έγινε χθε και στους δρόμους του Κιέβου και στα πλαίσια του Κοινοβουλίου, μέσα στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε επίση ότι η Ρωσική Δούμα σχεδόν ομόφωνα, 98% υπερψήφισε την απόφαση αυτή. Κατά την άποψή σας, ε, τι επίπτωση θα έχει αυτό στην κυριαρχία της Ουκρανίας και κύριε Επίτροπε μπορείτε να μας πείτε πώς θα επηρεάσει τις ε, ευρωπαϊκές προοπτικές της ε, Ουκρανίας και τις ευρωπαϊκές και τις ατλαντικές. Σίβιετς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην γνώμη σας για τη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Αυτή η συμφωνία δεν είναι μια συμφωνία όπου μια χώρα έχει ένα πλεονέκτημα και πληρώνει. Για 20 χρόνια υπήρξε μία άβυσος, ένα χάος. Για 20 χρόνια η Ουκρανία θα έχει φυσικό αέριο με χαμηλότερη τιμή και αυτά τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτό το φυσικό αέριο δηλαδή, δεν είναι λεφτά. Είναι έκπτωση. Δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία αγοράς ή μεταρρύθμιση της αγοράς. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το ρόλο της αντιπολίτευσης. Εμείς είδαμε ποια ήταν η κατάσταση χθες στο Κοινοβούλιο. Και, έγινε και ένα happening, ένα επεισόδιο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία. Και εγώ μίλησα με τον πρόεδρο Γιαννούκοβιτς. Και με όλο το establishment της ε, νέας εξουσίας. Μήπως είμαστε υπερισιόδοξοι. Η κυβέρνηση μπορεί να ακολουθεί τη δική της ε, πολιτική κυριαρχίας, αλλά μην ξεχνάμε τις άλλες προβληματικές. Κυρία Γιαντεμάκη για δύο λεπτά. χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Επισκέφτηκα και εγώ το ε, Νότιο Κάφκασο μόλις ε, πρόσφατα και διαπίστωσα ότι έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμως έχω ανησυχίες, τις εξής δύο. Πρώτη, το ορεινό Καραμπάχ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως περισσότερο, πιο ενεργά σε αυτό το θέμα. Τώρα ουσιαστικά ασχολούνται τα κλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι και τόσο ως ένωση. Γιατί είναι έτσι αυτή η κατάσταση και ποιο μέλλον διαβλέπετε εκεί, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τίποτα. Και ένα άλλο θέμα, το δεύτερο, θα έχει βουλευτικές εκλογές ε, προσεχώς το Αζερβαϊτζάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει θετικά εκεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να τη χώρα, αλλά γνωρίζουμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι πολύ αδύναμες όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξ όσων κατάλαβα, προσπαθούν να κάνουν δίκαιες και ελεύθερες εκλογές, αλλά χρειάζεται πολύ καιρό γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος η κυρία Ογιούλαντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις και μία ερώτηση προς την Επίτροπο. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωσή σας και για το έγγραφο το οποίο μας δώσατε. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με την συμφωνία της συνθήκη Χάρκοφα και εγώ ανησυχώ για τις επιπτώσεις της ε, συνθήκης αυτής ε, στο μέλλον. Από τη μια, ξέρουμε από την εμπειρία που έχουμε ότι το Κρεμλίνο μπορεί να αποσύρει να πάσα στιγμή την ε, συμφωνία του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι εγγυημένη παροχή φυσικού αερίου. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά την επιπτώσεις που θα έχει το ζήτημα αυτό στην ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και για την εξάρτηση που έχουμε για την ενέργεια μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα, όσον αφορά την διευκόλυνση των θεωρήσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου για το ζήτημα αυτό. Από τη δική μου εμπειρία γνωρίζω ότι και στην χώρα μου, την Εστονία, πριν από 10 χρόνια είχαμε θεωρήσεις για διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για, τον, για τους πολίτες της χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να θαρρύνουμε περισσότερο τη διαδικασία αυτή διευκόλυνση. Και κάτι ακόμα. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι θα συζητήσετε την ε, ιδιαίτερη εταιρική σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Θα μπορούσατε να μα πείτε περισσότερα πράγματα σχέση με αυτό. Σα ευχαριστώ. Προσετέθη μία τελευταία το, τοποθέτηση και είναι πραγματικά η τελευταία ογκουρεάνου λοιπόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφερθήκατε βεβαίως ε, θέματα θεώρησης ε, διαβατηρίων και άρση θεώρησης για χώρες που είναι στην πολιτική γειτονία. Φημολογείτε ότι θέλετε να δώσετε αυτό το καθεστώς πρώτα στη Ρωσία. Ισχύει αυτό ή είναι απλώς και δεύτερον, ε, ε, είπατε ότι το θέμα της Συμφωνίας Ουκρανίας-Ρωσίας είναι ε, θέμα διμερές, αλλά αυτό δεν ισχύει πάρα πολύ. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδιαφέρονται για την αντίληψή σας για τη συμφωνία αυτή και εσείς με τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Επίτροπος έχει το λόγο μέχρι και το πέρας της συνεδρίασής μας στις 12.30. Έχετε 9 τοποθετήσεις τις οποίες να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα ε, μέλη, ε, αγαπητέ κύριε Κύριλοφ, σε σχέση με το σχόλιο αυτό θα πρέπει να πω ότι η ε, ομάδα της οποίας είχα το προνόμιο να ηγούμε ήταν ακριβώς μια ομάδα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας σε στενή συνεργασία και με τη και τις υπηρεσίες της. Δηλαδή προσπαθήσαμε ήδη να εμφανιστούμε απέναντι στους συνομιλητές μας, όχι μόνο ε, κοινότητα, κοινοτική πολιτική, αλλά ε, και μετά τη Λισαβόνα, ε, την ΚΕΠΑ δηλαδή πολιτική. Σε σχέση με αυτά που ρώτησε ο κύριος Κυριλόφ για τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις από όλους τους βουλευτές. Η λογική εδώ ποια είναι. Νομίζω είναι σαφέστατη και απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν θέλουμε να παίξουμε σοβαρά ένα πιο παγκόσμιο ρόλο και να έχουμε μία φωνή στην εξωτερική πολιτική, θα έπρεπε ακριβώς να το διαμαδραματίσουμε αυτό το ρόλο. Και λυπάμαι, ε, συμφωνώ απολύτως με τη Βαρόνη ε, Άστον, ότι για να έχουμε παγκόσμια παρουσία θα πρέπει να αρχίσουμε από την κοντινή μας γειτονιά. Αυτό τι σημαίνει, ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε τα μέσα για να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο. Όχι βέβαια. Πολλές είναι οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες και σωστά συνδέεται και με την ε, ύπατη εκπρόσωπο κάθετο ε, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ούτε ίδια δεν έχει τα μέσα, ούτε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έτσι. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ε, είναι σε θέση και εκείνη να χρησιμοποιήσει πλήρως αυτό το μέσο και πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διαδραματίσει αυτό το μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα και βέβαια κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα. Και το Ορνό Καραμπάχ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ειδωθεί από τη σκοπιά των μέτρων ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Προσπαθούμε τώρα να στήσουμε μια πολιτική ε, στην Ένωση για κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας αυτή την υπηρεσία. Το ξέρουν και εκείνοι στην περιοχή. Μην περιμένετε λοιπόν θαύματα. Σιγά σιγά ε, θα ακολουθεί μια διαδικασία και στο τέλος θα ε, διαδραματίσει σημαντικότερο και μεγαλύτερο ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επίλυση της σύγκρουσης. Το 90% λέτε δεν αναφέρεται στη σύμβλεψή μας με την εξωτερική πολιτική. 90% των δηλώσεων και των δελτίων τύπου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούσα. Ε, έφεραν και την υπογραφή της Ουκρανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, ε, συμπαρατάσσεται κατά 90% μαζί μας. Και σε σχέση με τη συμφωνία για τη παράταση των βάσεων στη Σεβαστούπολη και τι σημαίνει αυτό θα το δούμε. Χρειάζονται πολλές αναλύσεις και εκτιμήσεις αυτού. Ο κύριος Στάλερ ρώτησε κάτι για τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις Γενέβης. Προσπάθησα να ξεκαθαρίσω ότι χρειαζόμαστε όχι απλώς να ε, συνεχίσουμε τις ε, συνομιλίες στη Γενέβη, αλλά και να τις επεκτείνουμε στο φάσμα τους, να μην καλύπτουν μόνο την πρόληψη επεισοδίου. Ανέφερα επίσης τη δυνατότητα της αποστολής μας στη Γεωργία ε, να εφαρμόζει πλήρως την εντολή της. Γνωρίζετε ότι αυτή είναι κατέρωθεν των ε, διοικητικών σύνορων η εντολή. Ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα. Ελπίζω να γίνει αυτό σύντομα. Ε, αυτό που έχει σημασία στο μεταξύ είναι η συνεργασία με τους Ρώσους με τρόπο που να πληρεί και η Ρωσία όλες τις ε, υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία Κατάπαυσης του πυρός, διότι δεν τις πλήρει ακόμα ε, εντελώς. Mr. Ε, κάποιος άλλος ρώτησε για το τι επίπτωση θα έχει αυτό στη διάσταση της ασφάλειας Πώς θα εξισορροπιστεί εκεί η κατάσταση και αυτό απομένει να καθαριστεί. Εμείς πήγαμε τη μεθεπομένη της ε, υπογραφής. Ας δούμε τι θα συμβεί. Έχω διαβεβαιώσεις του Προεδρού ότι, πώς να το πω, η αντιμετώπιση του θέματος αυτό με αυτόν τον τρόπο θα του επιτρέψει να δράσει καλύτερα και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η απόφαση για τις βάσεις δεν είναι έτσι παρόρμηση της στιγμής. Ανέλησαν τα σενάρια, τα ενδεχόμενα και την ε, λήξη ε, της Συμφωνίας για τις Βάσεις το 2017 της ενοικίασης. Ε, αυτά μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, η κυρία Αντρικένε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι από ό,τι φαίνεται οι Ρώσοι θέλουν ε, ε, παραπάνω από 25 ετία. Συζητούν για περαιτέρω παράταση δηλαδή. Βέβαια, ε, ξέρετε ότι η βάση είναι εκεί χρόνια ολόκληρα τώρα, δεν είναι πρόσφατη και τι θα σημαίνει αυτό για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το είπα και στο Κίεβο. Ε, θα κριθούν από τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους. Και όχι από το αν θα ε, υπάρχει στρατιωτική βάση των Ρώσων εκεί. Για τον κύριο Σίβιτς, για μας είναι σημαντικό και ήταν σημαντικό να μας διαβεβαιώσουν οι Ουκρανοί ότι πρώτον η συμφωνία αυτή δεν σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα ε, προχωρήσει ε, στην εισαγωγή ε, ευρωπαϊκών τιμών για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Έτσι. Και επίσης ότι δεν θα επηρεάσει τις κοινέ μας δράσεις και σχέδια να εξυγχρονίσουμε το σύστημα των αγωγών που διέρχονται μέσω της Ουκρανίας. Και μας διαβεβαίωσαν ότι όχι, όχι, εντάξει, μας καθυσίχασαν. Optimism. I think, uh, ε, για την αισιοδοξία. Εγώ το ξεκαθάρισα. Σε τελική ανάλυση, η δική μας η ε, αισιοδοξία δεν ε, θα βασιστεί ούτε θα κριθεί από τα λόγια και τις υποσχέσεις και τα όσα ε, μαστάζουν οι Ουκρανοί, αλλά τα όσα θα έχουν κάνει. Και αυτό που είχε σημασία ήταν να τους δώσουμε να καταλάβουν και να καταλάβουν και εμείς ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία θα πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη. Και ένα δεύτερο στάδιο. Χρησιμοποιούμε αυτή τη μήτρα από το Matrix και ε, τη ε, διαδικασία για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και στο Κίβο είπε κάποιος διπλωμάτης πολύ χαρακτηριστικά Από λόγια καλά τα πάνε. Για να δούμε τώρα στη πράξη τι θα κάνουν. Βέβαια δεν είναι δική μου αυτή η παράθεση έτσι. Η κυρία Γιατεμάκη ρώτησε για τον Αγκόνο Καραμπάχ. Νομίζω ότι απάντησα ήδη σε αυτό. And I, hope that uh, by the time... Και ελπίζω να διαδραματίσει πραγματικά πιο ενεργό και θετικό ρόλο η Ένωση. Ο Γιούλαντ. Η κυρία Γιούλαντ ρώτησε. Μήπως αποσύρει η Ρωσία την υπογραφή της. Μα κοιτάξτε, δεν έχουμε δύο διαφορετικές συμφωνίες. Δεν έχω φέρει το κείμενο μαζί μου, το ρωσικό που μου έδωσαν τη συμφωνία. Δισέλιδο είναι. Με μία υπογραφή και μόνο. Αυτές οι δύο σελίδες αφορούν και τη συμφωνία για το φυσικό αέριο αλλά και για τη στρατιωτική βάση. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα διαχωριστούν. Δεν είναι δύο ξεχωριστές συμφωνίες. Είναι στην ίδια συμφωνία συνδέονται και τα δύο ζητήματα. Σημασία είχε για τις Ουκρανικές αρχές να καταργηθεί ε, αυτή η συμφωνία του περασμένου Ιανουαρίου, του περσινού. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω καθόλου τη θέση τους, όχι, ε, σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είχαν και πολλά μέσα στη διάθεσή τους. Ένα από τα μέσα που είχαν ήταν να κάνουν τη Ρωσία να ενδιαφερθεί και να συμμετέχει στο σύστημα διαμετακόμισης του φυσικού αερίου. Όπως γνωρίζετε, ε, η Ρωσία όμως φτιάχνει ε, αγωγούς North Stream και, North, ε, και South Stream. Δηλαδή κάνουν ό,τι μπορούν για να παρακάμψουν. Να μην είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το σύστημα διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας. Δηλαδή, οι Ουκρανοί δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο. Και δεν έχουν και πάρα πολλές άλλες συναλλακτικές λύσεις στα χέρια τους επαναλαμβάνω και πάλι τι εξηγήσει που μα έδωσαν. Δεν σημαίνει ότι του υπερασπίζομαι. Ούτε είναι θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου. A special partnership with, with Azerbaijan. Η ειδική σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Δεν είναι μέλο του ΠΟΕ το Αζερβαϊτζάν. Uh, uh, ε, σε εκείνο εναπόκειται να πάρει την απόφαση εάν θα ενταχθεί ή όχι. Και πότε. Εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, ότι δεν είναι ακριβώς στην αυριανή ημερήσια διάταξη αυτό. Δηλαδή, δεν είναι του παρόντος, δεν πρόκειται να κάνει ε, αυτή τη διαπραγμάτευση ε, προκειμένου με την Αρμενία. Αυτό θα μας ε, δυσκόλευε και τα πράγματα για μας ε, και είμαστε σε εντατικές ε, συσκέψεις και με τους εταίρους μας εκεί και τελικά καταλήξαμε να προτείνουμε το εξή. Ας ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία προσχώρησης, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η εντολή είναι αρκετά ευέλικτη για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακόμα και χωρίς παράλληλη έναρξη ε, ε συνεργασία για την οικονομική ολοκλήρωση και στο ε, μεταξύ παραλλήλως να μεγιστοποιήσουμε τι συμφωνίες που έχουμε τώρα, οι συμβατικές υποχρεώσεις με το Αζερβαϊτζάν υπό την παρούσα μορφή. Έχουμε μια σειρά ε, δυνατοτήτων ευθυγράμμισης του Αζερβαϊτζάν σε πολλές από τις δικές μας εσωτερικές πολιτικές. Έτσι. Uh, Στη συνέχεια, εκφράστηκε επιθυμία σαφής εκατέρωθεν να ξεπεράσουμε ε, το, ενεργειακό τομέα. Να μην συζητούμε μόνο αυτό, όχι να τον αγνοήσουμε καθόλου, αλλά να ε, αντλήσουμε πλεονεκτήματα από την ενέργεια, γιατί είναι κινητήρια δύναμη όχι μόνο εξυγχρονισμού της ίδιας της χώρας του Αζερβαϊτζάν και όσοι έχετε πάει πρόσφατα στο Αζερβαϊτζάν θα το επιβεβαιώσετε αυτό. Το βλέπετε μπροστά στα μάτια σας να αλλάζει. Αλλά είναι και κινητήρια δύναμη για πιο ευρεία βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξυγχρονιστεί η κοινωνία του Αζερβαϊτζάν και συνολική, επαναλαμβάνω. Γιατί όταν αναφαθμίζεις την οικονομία σου, το κοινωνικό σύστημα, ε, όχι κατά ένα επίπεδο, αλλά ένα, και ένα και δύο και τρία επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσεις και άλλα θέματα, δεν είναι αυτόματα, και την παιδεία, αλλιώς... Ε, αργά ή γρήγορα αντιμετωπίζουν προβλήματα οι κοινωνίες, εάν ποντάρουν μόνο στην οικονομία και με ταχύ ρυθμού ε, αναπτύσσονται. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα, Γι' αυτό μιλώ για μια ειδική εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ήδη από τώρα κάποιες πρώτες ιδέες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, θα επισκεφθεί το Αζερβαϊτζάν. Κατά αυτόν τον τρόπο θα, να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε καλύτερα τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα ανάμεσα στον πρόεδρο της χώρας και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Γκεριάνο για τις θεωρήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. ξέρω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική για το τι απαιτείται να γίνει στα πλαίσια του απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και θεωρούμε ότι εδώ θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη που έχουμε χρησιμοποιήσει και για τα Βαλκάνια. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή για την Ουκρανία μιλάμε για έναν οδικό χάρτη, για μια προσέγγιση οδικού χάρτη όσον αφορά τις θεωρήσεις. Οι συζητήσεις όμως ακόμα θα πρέπει να γίνουν και κυρίως από τους Υπουργούς Εσωτερικών. Και μολονότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να πάρουν την απόφαση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα προσεγγίσουμε το πολύ πολιτικά ευαίσθητο αυτό ζήτημα και πολύπλοκο από τεχνικής πλευράς με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά από ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν λαμβάνοντας απλώς υπόψη μας κάποιες πολιτικές εκτιμήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις πολύ καλές, πλήρεις, διεξοδικές απαντήσεις που μας έδωσε και για τη διεξοδική ενημέρωση που μας έκανε στην αρχή. Ξεκινήσαμε πολύ καλά τη συνεργασία μας και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί ακόμα καλύτερη συνεργασία μας, κύριε Επίτροπε, στο μέλλον. Η επόμενη συνάντησή μας με τον Επίτροπο θα λάβει χώρα στις 17 Μαΐου στο Στρασβούργο και θα ενημερωθούμε τότε περισσότερο για κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας, για την εργό συμμετοχή σας. Θα συνεχίσουμε πάλι στις 3 η ώρα με τον κύριο Προβέρα στην Προεδρία. Σας ευχαριστώ.